Καλημέρα σε όλους αγαπητοί συνάδελφοι. Σας καλωσορίζω στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής μας ε, το 2018. Ελπίζω να είχατε όλοι ένα ευχάριστο διάλειμμα στις διακοπές των Χριστουγέννων και ελπίζω να συνεχιστεί η καλή μας συνεργασία στην Επιτροπή μας ε, κατά τους επόμενους 6 ε, μήνες ή μάλλον συγγνώμη 12 μήνες. Περνάω στο πρώτο σημείο έγκριση τη σα διάταξη. Δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσει, οπότε εγκρίνεται. Δεύτερον, σημείο ανακοινώσει του Προέδρου. Δεν έχω κάτι να ανακοινώσω, οπότε περνάμε κατευθείαν στο σημείο 3, έγκριση δηλαδή των πρακτικών των συνεδριάσεων τη Δευτέρα Οκτωβρίου, τη 9η και 10η Οκτωβρίου, τη 19η Οκτωβρίου, τη 23η Οκτωβρίου και τη 6η Νοεμβρίου. Αν δεν υπάρχουν λοιπόν σχόλια σε σχέση με αυτά τα πρακτικά έω το πέρα τη συνεδρίαση, θα θεωρηθούν εγκεκριμένα. Περνάμε λοιπόν κατευθείαν στι ψηφοφορίε και νομίζω πως θα χρειαστούμε τουλάχιστον μία ώρα για να ολοκληρώσουμε όλες αυτές τις ψηφοφορίες και ξεκινάμε με την πρώτη από αυτές τις ε, ψηφοφορίες, δηλαδή τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία με συντάκτη αυτή τη νομοδότηση τον συνάδελφο Μαμίκιν. Δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι, Αντρές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ τους κοιόδες συζητητές για τη συνεργασία που είχαμε, τους κοιόδες συζητητές, συγγνώμη, και ελπίζω να υπάρξει μεγάλη συνένεση στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Ε, δεν βλέπω να υπάρχουν σχόλια, οπότε α περάσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία.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 την ελέγχουμε. Ελέγχουμε λοιπόν τη 48. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Απορρίπτεται λοιπόν. 50 υπέρ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 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε την 62 άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 36 πέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και περνάμε στην ψηφοφορία επί του συνόλου της νομοδότησης. Τελική λοιπόν ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέραση ψηφοφορία ψηφοφορίας. Και εγκρίνεται με 48 ψήφους υπέρ και 3 κατά. Περνάμε στο σημείο 5, το επόμενο δηλαδή πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, προετοιμασία τη θέση του Κοινοβουλίου για το επόμενο πλαίσιο μετά το 2020. Ο συντάκτη ε, τη νομοδότηση είναι ο κ. Παντζέλη, δεν ξέρω αν θέλει να πάρει το λόγο. Όχι, καλώ, μπορούμε να περάσουμε κατευθείαν στη πληροφορία. Ξεκινάμε λοιπόν με την συμβιβαστική τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 24. Τμήματική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα, ένα C δηλαδή υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική τροπολογία 1 Ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρα τη ψηφοφορία, αφού ψήφισαν όλοι, απορρίπτεται λοιπόν με 41 ψήφου κατά και 3 υπέρ. Οπότε περνάμε στην προφορική τροπολογία υπαριθμών 2. Και πάλι εδώ ονομαστική ψηφοφορία. is disclosed, that has been rejected. Πέραση εφορία. Απορρίπτεται λοιπόν. Προφορική τροπολογία 3. Ονομαστική και πάλι ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται λοιπόν. Περνάμε τώρα στην βασική τροπολογία 5. Περ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές. Ας ελέγξουμε τη συμβαστική τροπολογία 11, άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Απορρίπτεται λοιπόν τη συμβαστική τροπολογία 11 με διαφορά μιας ψήφου. Οπότε περνάμε στην 47 επέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ας την ελέγξουμε. Ας ελέγξουμε λοιπόν την τροπολογία 47 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Α, καταπίπτει, ζητά συγγνώμη ο πρόεδρος. Καταπίπτει η 47 γιατί εγκρίθηκε η συμβαστική τροπολογία 6. Άρα περνάμε στην τοπολογία 51. τοπολογία 51 λοιπόν. Υπέρ, κατά, αποχές. So that was rejected. Απορρίφθηκε λοιπόν και περνάμε στην 63. Υπέρ, κατά, αποχές. Ας ελέγξουμε την 63. Είπε, Είμαστε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται λοιπόν η 63. Περνάμε τώρα στην ηλεκτρονική ψηφοφορία επί του συνόλου της νομοδότησης. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρασε τη ψηφοφορία λοιπόν και εγκρίνεται η γνωμοδότηση. Και φτάνουμε στο σημείο 6. Uh, the result was 39-4-9 again. Είχαμε 39 υπέρ, 9 κατά και μερικές αποχές. Λοιπόν, 6. Απαλλαγή 2016, Γενικός Προϋπολογισμός, ε, ΕΙΕΔ. Ο κύριος Πρέντα είναι ο εισηγητής, ο οποίος φαίνεται ότι δεν είναι εδώ σήμερα. Θα ήθελε κάποιος άλλος να λάβει το λόγο, φαίνεται πως όχι. Άρα περνάμε στην ψηφοφορία. Amendment number one. Ένα υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία υπαριθμών 1 έλεγχος. It's closed. Πέρας. Εγκρίθηκε 28 έναντι 24 ψήφων. Δύο υπέρ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 9. Τμηματική ψηφοφορία. Α, καταπίπτει γιατί εγκρίθηκε η 8. Όχι, δεν εγκρίθηκε η 8. 9 λοιπόν, υπέρ. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εγκρίθηκε το 9, ναι. 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 14 ξεχωριστή ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 16 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά το προσχέδιο όπως τροποποιήθηκε, άρχεται η ψηφοφορία. It's closed. Πέρας. Εγκρίνεται 49 έναντι 6 ψήφων. Και τώρα ψηφίσουμε το 7 απαλλαγή 16 Γενικός Προϋπολογισμός Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Πρέντα είναι εισηγητής. Ο κύριος Παντσέρη όμως θα ήθελε να λάβει το λόγο, ο οποίος και τον έχει. Ήθελα απλώς να προτείνω μία προφορική τροπολογία στην 17 του κυρίου Σολέ. Δεν ξέρω αν θέλετε να την αναφέρω τώρα ή να περιμένω να φτάσουμε στην 17. Θα ήθελα να διαγραφεί ένα μέρος αυτού του, ε, αυτής της τροποποίησης, ως προφορική βεβαίως, που προτείνω τώρα. Όταν φτάσουμε στην 17. Εντάξει. Άλλα σχόλια. Μπορούμε λοιπόν να αρχίσουμε την ψηφοφορία μας. 1 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ. Κατά αποχές. Ας ελέγξουμε την 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 7 με την προφορική 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 Κύριε Πανζέρη, σας ακούμε. Ήθελα να διαγράψουμε το δεύτερο τμήμα αυτής της τροπολογίας. Δηλαδή εκφράζει την ανησυχία μέχρι το Ισραηλινές αρχές και να διαγράψουμε αυτό που λέει ότι ζητάμε από την Επιτροπή να μειώσει μέχρι για το Ισραήλ. Δηλαδή το δεύτερο τμήμα να διαγραφεί. Είναι σαφές. Αυτό είναι το αίτημα του κυρίου Παντζέρη, λοιπόν. Ποιος αντιτίθεται. Αρκεί ένα. Τέσσερις συνάδελφοι είναι κατά, άρα απορρίπτεται κύριε Παντζέρη η προφορική. Το αίτημα προφορικής. Ψηφίζουμε την 17 ως έχει, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και φτάνουμε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία της ε, ε, τροποποιημένης έκθεσης. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 50 έναντι 3. εφαρμογή του κοινού εγγράφου εργασίας, ισότητα των φύλων, αλλάζοντας τη ζωή των κοριτσιών και των γυναικών. Η κυρία Μπεατρίθ Μπεθέρα Μπασταρετσέα είναι η συγγήτρια. είναι παρούσα. Φαίνεται πως όχι. Θα ήθελε κάποιος να λάβει το λόγο. Miss would you like to... Κυρία Μπασταρετσέα, θα θέλατε να πείτε κάτι. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις για αυτή την έκθεση. Ήταν μεγάλη χαρά να συνεργαστώ μαζί τους και θα θέλαμε να συνεισφέρουμε σε αυτόν τον ε, κοινό στόχο, δηλαδή την αλλαγή της ζωής των κοριτσιών και των γυναικών. Κάποιος άλλος? Φαίνεται πως όχι. Άρα περνάμε στην ψηφοφορία. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται.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 πέρας εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 61 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά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 Εγκρίνεται 53 ψήφοι έναντι 5. Και περνάμε λοιπόν τώρα στο σημείο υπαριθμών 9, δημιουργία του Ευρωπαϊκού Προγράμματο Βιομηχανική Ανάπτυξη στον τομέα τη άμυνα με σκοπό την στήριξη τη ανταγωνιστικότητα και τη ικανότητα κοινοτομία τη αμυντική βιομηχανία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρξαν κάποιε συζητήσει ε, από ό,τι ενημερώθηκα και θα ήθελα να δώσω λοιπόν το λόγο πρώτα. ποιο ε, θέλει να πάρει το λόγο, ο κύριος Γιουρέκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν να περάσουμε στην ψηφοφορία, θα ήθελα να δηλώσω το εξή. Στην τελευταία έκθεση θα α, θέσω ένα ξεχωριστό ερώτημα στην προηγούμενη έκθεση. Στην προηγούμενη έκθεση, διευκρινίζει ο Πρόεδρος. Ναι, για την προηγούμενη έκθεση. Στην τελευταία, την προηγούμενη έκθεση, την οποία μόλις ψηφίσαμε. Το ανακοινώνω απλά. Okay. So, can we go back now to item number nine? Μάλιστα, ας περάσουμε στο σημείο υπαριθμών 9 πάλι. Ο κύριος Πάσκου είναι ο εισηγητής. Θα θέλει κανείς να πάρει το λόγο, ο εισηγητής μήπως. Όχι. Ποιος θα θέλει να πάρει το λόγο, παρακαλώ. Ο κύριος Καστάλτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφέρω ως προς την έκθεση Πάσκου ότι είχαμε ε, αιτήματα για αναβολή της ψηφοφορίας γιατί δεν συμφωνήσαμε σε ένα βασικό σημείο. Από τις ανταλλαγές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ελέγχθη ότι θα πρέπει να αναβληθεί για αργότερα, απόψε δηλαδή, γιατί πολλοί δεν έχουν καν τον κατάλογο μπροστά τους. Θα θέλαμε λοιπόν να αναβληθεί ή αργότερα ή για την 1η Φεβρουαρίου, αλλά ίσως αργότερα σήμερα. Σας ευχαριστώ κύριε Καστάλτο. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. κυρία Βαλέρο. Ήθελα απλά να συμφωνήσω απόλυτα 100% με τον κύριο Καστάλτο. Νομίζω ότι δεν είχαμε το σωστό χρόνο να κοιτάξουμε τις τροπολογίες και άρα θα χρειαστεί αναβολή. Εγώ θα προτιμούσα για το Φεβρουάριο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στη χειρότερη περίπτωση για το απόγευμα. Ευχαριστώ, κύριε Βαλέρο, Λέει ο πρόεδρος, ο συνάδελφος από τους Βιλελευθέρους, ο κύριος Ραντός. Η Άλντε επίσης θα ήθελε να υποστηρίξει την πρόταση αυτή που έγινε. Μάλιστα, ευχαριστώ κύριε Τανζό. Κοιτάξτε, εμεί είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε εδώ τώρα το πρωί. Καταλαβαίνω τι ζητούν οι συνάδελφοι που ζητούν αναβολή για σήμερα το απόγευμα, αλλά θεωρώ ότι είναι λίγε οι τροπολογίες που είναι αμφιλεγόμενες. Άρα θεωρώ ότι μπορούμε να τις λύσουμε. Γι' αυτό λοιπόν δεν θέλαμε να γίνει αναβολή για τον Φεβρουάριο. Ε, για μας να γίνει η ψηφοφορία το συντομότερο δυνατόν, τώρα, σήμερα. Και ζητώ να συμφωνήσουμε, παρακαλώ. Μάλιστα, κύριε Σπάσκο, τι λέει. Εγώ συμφωνώ. Συμφωνώ ήταν πάρα πολύ σφιχτό το χρονοδιάγραμμα, αλλά από ό,τι κατάλαβα η πρωτοβουλία εξαρτάται και από το χρονοδιάγραμμα αυτό. Νομίζω ότι ξέρουμε ότι μία μικρή αναβολή μέχρι το απόγευμα δεν θα βλάψει το γενικότερο χρονοδιάγραμμα. Θα πάρει η ΙΤΡΕ, η Επιτροπή Βιομηχανίας, την γραμμοδότησή μας στην ώρα της. Ε, άρα αυτό το δέχομαι. Το μόνο πρόβλημα είναι το εξής αν ψηφίσουμε στην αρχή του απογεύματος, το μεσημέρι δηλαδή και μετά, ή λίγο πιο μετά, στο τέλος του απογεύματος, γιατί ενδεχομένως κάποιοι συνάδελφοι να μην έχουν προβλέψει να είναι παρόντες και να έχουν άλλες υποχρεώσεις. Άρα εδώ θα πρέπει να δούμε στις τρεις μας κάνει ε, ο πρόεδρος. Ε, συνάδελφοι, να κάνω μια πρόταση. Σήμερα το απόγευμα θα γίνει ένα debriefing για την ε, στις 2.30 για την αποστολή μας στο Νίγηρα. Προτείνω λοιπόν να ψηφίσουμε στις 2.30 και μετά να γίνει το debriefing η ενημέρωση, δηλαδή ακριβώς μετά την ψηφοφορία. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη δυνατή λύση αυτή. Στις 2.30 λοιπόν το απόγευμα συμφωνούν όλες οι πολιτικές ομάδες. Παρακαλώ για την αναβολή αυτή. Μάλιστα. Άρα το σημείο 9 αναβάλλεται. Η ψηφοφορία θα γίνει στις 2.30 το απόγευμα, σήμερα το απόγευμα. So we are through... Έτσι λοιπόν ολοκληρώσαμε τις πιο πολλές ψηφοφορίες που είχαμε για σήμερα. Ο κύριος Νάρτ είναι εδώ παρακαλώ. Gracias, señor presidente. No, not yet. Wait a moment. Όχι, όχι, περιμένετε. Colleagues, could you please... Συνάδελφοι, σας παρακαλώ, αν δεν θέλετε να συμμετέχετε στην συζήτηση για το επόμενο θέμα, παρακαλώ, συνάδελφοι, βγείτε από την αίθουσα. Wieso? Now, item number 10. Να περάσουμε στο σημείο 10, λέει ο Πρόεδρο. Σύσταση προ το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση σχετικά με την εξάλληψη των πηγών εσόδων των τσιχαντιστών. Στόχο θετημένη καταπολέμηση τη χρηματοδότηση τη τρομοκρατία. Και ο Χαβιέ Νάρτ είναι ο εισηγητή μα. Ε, με ενημέρωσαν ότι η συνάντηση των σκιωδών ήταν πάρα πολύ παραγωγική και καταλήξαμε σε μια συμφωνία για τι συμβαστικέ τροπολογίε. Οπότε και δίνουμε το λόγο στον κύριο Νάρτ. Είναι μια σύσταση πολύ σημαντική γιατί πρόκειται για την χρηματοδότηση, την τρέχουσα χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Ε, ως προς μία Χρηματοδότηση που είχε αρχίσει με τους δίδυμους πύργους. Τώρα περνάμε όμως σε μικροχρηματοδότηση που μπορεί να δημιουργήσει τεράστιες ε, τραγωδίες όπως της Νίκιας ή της Βαρκελόνης που πραγματοποιήθηκαν με πενιχρά οικονομικά μέσα. Γι' αυτό έγιναν ε, μεγάλες μεταφορές χρημάτων στο παρελθόν, αλλά τώρα δεν γίνονται τόσο μαζικές μεταφορές ε, τραπεζικής, ε, τραπεζικές μεταφορές χρημάτων. Γι' αυτό μας ενδιαφέρει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ελέγξουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την μικροχρηματοδότηση και φυσικά θα πρέπει να υπάρξει προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτό αποτελεί πρόκριμα αυτής ε, της σύστασης για να υπάρξει μία υποστήριξη ε, σε... και υλοποίηση ενός σχεδίου κατά της Ισλαμοφοβίας. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι απολύτως αναγκαίο να δημιουργηθεί μία πλατφόρμα όπου οι υπηρεσίες πληροφοριών των κρατών μελών να μπορέσουν να έχουν ένα σταθερό τόπο για μεταφορές πληροφοριών. Και αυτό για έναν λόγο, για να μην δημιουργήσουμε μία, ένα νέο κέντρο και μία νέα οργάνωση, γιατί ε, είναι αντιπαραγωγικό. Οι υπηρεσίες πληροφοριών κινούνται στα πλαίσια εμπιστοσύνης. Γι' αυτό το να δημιουργήσουμε ένα θεσμικό όργανο, να θεσμοθετήσουμε αυτό το πλαίσιο, δεν θα ήταν σκόπιμο. Θα πρέπει να είμαστε πραγματιστές και πρακτική. Δεύτερον, θα πρέπει να ελέγξουμε τις μικρομεταφορές, ιδιαίτερα εκείνες μέσω των παραδοσιακών κυκλωμάτων από την Χαουάλα της Αραβίας μέχρι την Πάταλα το που είναι ένα σύστημα στις Φιλιππίνες. Οποιοδήποτε δηλαδή σύστημα μικρομεταφορών εκτός γνωστών κυκλωμάτων. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να υπάρχουν ε, διακρίσεις γιατί μπορεί κανείς να ανήκει σε μια εθνική πολιτιστική ομάδα που να ακολουθεί διαφορετικές μεθόδους από τους συμπατριώτες του. Εάν λοιπόν μπορεί να υπάρχει έλεγχος των μεταφορών από τα προϋπάρχοντα συστήματα, είναι σκόπιμος. Επίσης, η επαναφόρτιση των καρτών γίνεται μέσω ενός συστήματος ελέγχου από τον λογαριασμό όψεως ή από άλλους λογαριασμούς. Συμφωνήσαμε λοιπόν για τον έλεγχο αυτών των ε, καρτών και επίσης ε, τη χρηματοδότηση μέσω ενιαίου νομίσματος. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τις θρησκευτικέ οργανώσεις ή τις πολιτιστικές οργανώσεις που την χάνουν αυτού του είδους χρηματοδότησης. Υπάρχουν, υπάρχουν και τα κρυπτονομίσματα όπως το bitcoin και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να προτείνουμε στην Επιτροπή ένα ε, συγκεκριμένο ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο να μπορεί να υλοποιηθεί. Και πιστεύω ότι οι 281 τροπολογίες που λάβαμε ήταν πολύ σημαντικές καθώς και η δράση των διαφόρων ομάδων που αποτελεί μία απτή πραγματικότητα. Γι' αυτό υπήρξε συνένεση με μεγάλη πλειοψηφία ως προς μία πρόταση της Επιτροπής και όλες ε, οι ομάδες γνωρίζουν τις άμεσες, άμεσες ανάγκες μας. Είμαστε πραγματιστές και γι' αυτό θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους εμπλεκόμενους και τις πολιτικές ομάδες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Νάρτ. Και τώρα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση από πλευρά της, ε, του ΕΛΚ. Ο κ. Ντάκτουσον, ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα να ξεκινήσω σχολιάζοντας αυτά που είπε ο κύριος Νάρτ και ε, δίνοντα ε, συγχαρητήρια στον κύριο Νάρτ, γιατί ήταν πραγματικά πολύ επικοδομητικέ οι διαπραγματεύσει. Συμπεριλήφθηκαν και πολλέ από τι τροπολογίε που ήταν σημαντικέ για μα, για το ΕΛΚΑ. Να αναφέρω λοιπόν κάποιες από τις προτεραιότητες για την ομάδα μας σε ό,τι αφορά το τραπέζι των διαπραγματεύσεων στην 11, ε, την συμβαστική 11. Θέλαμε να τονίσουμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο και να θεωρήσουν με βασική πολιτική της προτεραιότητα τη μείωση και την εξάλληψη των εισόδων για τέτοιες οργανώσεις. Και υπάρχει η πλατφόρμα για την τρομοκρατία, ενώ παράλληλα θέλουμε να υπάρξει και μία διευκρίνηση ότι αυτό δεν θα πρέπει να σημαίνει ότι θέλουμε να δημιουργηθεί άλλη μία υπηρεσία. Η Συμβαστική 13 τώρα για την Ομάδα Εργασίας για την Οικονομική Δράση. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι το σώμα αυτό ανέπτυξε μία στρατηγική για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και μας ικανοποιεί η συμπερίληψη του συντονιστή για την τρομοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 19 Συμβαστική Τροπολογία για να έχει ένα ρόλο στην κατάρτιση του καταλόγου για τις οργανώσεις και τα άτομα τα οποία λειτουργούν υπό μη διαφανή καθεστώτα. Το γεγονός ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει ζητήσει από την διεθνή κοινότητα να αυξήσει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης τη τρομοκρατία, αναφέρεται στην τροπολογία υπαριθμών 20. Είμαστε σύμφωνοι. Και στην τροπολογία 21 τώρα, τη συμβιβαστική. Υπήρχαν διαφορετικέ απόψει για το κατά πόσον το αρχικό κείμενο το οποίο αναφέρει τι μάσκε θα πρέπει να παραμείνει ή όχι. Η πιο πολλοί ήταν υπέρ τη διαγραφή. Εγώ Χρειάστηκε να μιλήσω και με τους συναδέλφους, γιατί το ΕΛΚ υποστηρίζει την εποπτεία από τις αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της χρηματοδότησης από ξένες, ο, συγγνώμη, όχι για μάσκες, αλλά για τζαμιά, τη χρηματοδότηση για, την, για τα τζαμιά. Και πιστεύουμε ότι η χρηματοδότηση τέτοιων θα μπορούσε να αυξήσει την τρομοκρατία και τις τρομοκρατικές δράσεις ε, στις χώρες μας. Και θα ήθελα κλείνοντας να αναφέρω τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εστιαστεί σε κάποιες δομές προτεραιότητας η απάντηση στο ερώτημα του κατά πόσο χρειάζεται πιο πολύ ή πιο λίγη ευρωπαϊκή συνεργασία είναι τι Και τα δύο χρειάζονται. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την λήψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Από τη φύση της άλλωστε η τρομοκρατία δεν γνωρίζει σύνορα. Ενώ και τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία είναι τα πλέον αρμόδια να λαμβάνουν αποφάσεις για θέματα όπως για παράδειγμα κοινωνική πολιτική. Να σας πω ότι υπάρχει και χαίρομαι που υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία υπέρ της ε, προσπάθειας αυτής η οποία χρειάζεται διεθνή συντονισμό. Με τις κοινές αυτές προσπάθειες η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να το επεξέλθει. σε ό,τι αφορά δηλαδή το κεφάλαιο που θρέφει τους τζιχαντιστές. Η έκθεση είναι καλογραμμένη, ισόρροπη κύριε Πρόεδρε και νομίζω ότι συμβάλλει προς το στόχο μας, τον οποίο ασφαλώς και υποστηρίζω. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Αντάκτουσον. Για σοσιαλιστές τώρα, Κλέρ Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την επικοδομητική του συνεργασία με όλους μας σε σχέση με αυτό το φάκελο. Ε, υπήρξαν ε, καλοί συμβασμοί στους οποίους καταλήξαμε συμπεριλαμβανομένων των τροπολογιών ε, σε σχέση με το Financial ε, Action Task Force και αυτή την πρόταση σε ό,τι αφορά τη δημιουργία μιας νέας πλατφόρμας η οποία όμως θα βασίζεται σε υφιστάμενες δομές. Ε, η πλατφόρμα λοιπόν αποτελεί μια καλή ιδέα ε, προκειμένου να έχουμε μια καλύτερη αντίληψη του κινδύνου τον οποίο αντιμετωπίζουμε. Επίσης θα ήθελα να ε, χαιρετήσω εδώ την εσκεμμένη προσπάθεια που κάνει ο εισηγητής να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα με αποτελεσματικό τρόπο. Και τον ευχαριστώ για τη συνεργασία του σε σχέση με αυτό το ζήτημα με τους εστιώδεις εισηγητέ, ε, προκειμένου να τοποθετηθούμε λεπτομέρως σε σχέση με αυτό. Όμως ε, για να αποφύγουμε ε, μια Ισλαμοφοβία και προκειμένου να εστιάσουμε σε πραγματικά απτά αποτελέσματα και την αντιμετώπιση του προβλήματος στην πηγή του, δεν χρειάζεται να προβαίνουμε σε εμπριστικές δηλώσεις. Με βάση λοιπόν τις συζητήσεις ε, που έγιναν και με βάση την ε, πολύ καλή δουλειά που κάναμε από κοινού, αναμένω πω η τελική εκδοχή του κειμένου θα είναι ε, πραγματικά ρεαλιστική ω προ τι προτάσει που θα κάνει σε σχέση με την ανταλλαγή πληροφοριών και την αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της δημοκρατίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος την Τώρα για το ECR δεν βλέπω να ζητά σε το λόγο. Κυρία Σακοράφα λοιπόν τώρα για την κουρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Νάρτ για την σημαντική προσπάθεια που έκανε για να μας παρουσιάσει μια συμπεριληπτική και ισορροπημένη έκθεση. Θεωρώ ότι η απάντηση στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας δεν μπορεί να είναι μονοδιάστατη και φυσικά δεν πρέπει να εστιάζεται μονάχα στην αποτροπή των τρομακρατών από την χρήση του διεθνού χρηματοπιστωτικού συστήματο, που κακά τα ψέματα κύριε συνάδελφοι είναι το ίδιο που αναπτύσσει και υιοθετεί όλα τα μέσα που χρησιμοποιούν οι τρομοκράτε για την χρηματοδότησή του. Η πραγματικότητα έχει δείξει ότι αυτό ο προσανατολισμό είναι υποκριτικό, αφού σήμερα οι περισσότερε επιθέσει που καταγράφονται ειδικά στην Ευρώπη απαιτούν πολύ λίγα χρήματα και οι τρομοκράτε χρησιμοποιούν ένα μεγάλο φάσμα αποτελεσματικών μεθόδων μεταφορά χρημάτων και συγκέντρωση κεφαλαίων όταν χρειάζεται να αποφεύγουν το διεθνέ χρηματοπιστωτικό σύστημα. Έχουν περάσει 19 χρόνια από το πρώτο σχετικό ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών. Δρούν σήμερα περισσότερε τρομοκρατικέ οργανώσει με περισσότερα χρήματα από ποτέ άλλοτε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να εστιάσει σε δύο επίπεδα σε πολιτικό επίπεδο θα πρέπει να μας πει ποια κράτη ή καθεστώτα κρατών με τα οποία συνεργάζεται έχουν συμμετάσχει είτε άμεσα είτε έμεσα με την ανοχή του στη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων. Τον ΤΑΕΣ γνωρίζουμε ότι αποτελεί μονάχα ένα παράδειγμα και θεωρώ είναι υποκριτικό να προσποιούμαστε ότι προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία συνεργαζόμενοι με χώρες που εσκεμμένα επιτρέπουν την εκόλαψή τους. Όσον αφορά το τεχνικό επίπεδο, το, σε αυτό το κομμάτι το ψήφισμα αναφέρει πάρα πολλά, τα ανέφερε και ο κύριος Νάρτ, δεν θέλω να τα ανασταθώ σε αυτά. Θα πρέπει όμως ε, να σέβονται πλήρως τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, τα προσωπικά δεδομένα και τον σεβασμό κυρίως της ιδιωτικής ζωής. Τελικά, αν θέλει πράγματι η Ευρωπαϊκή Ένωση να απαντήσει στο ζήτημα της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, θα πρέπει να αναλάβει διεθνείς πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των παράνομων οικονομικών δομών σε περιοχές που αναπτύσσονται τρομοκρατικές οργανώσεις. Από αυτή την άποψη, η προώθηση της ανάπτυξης, η βελτίωση της διακυβέρνησης και η καταπολέμηση της διαφθοράς μπορούν να παίξουν σημαντικότερο ρόλο από την αποτροπή των τρομοκρατών από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Και φυσικά θεωρώ πολύ σημαντική προς αυτή την κατεύθυνση την αναφορά στην ανάγκη να μπει ένα τέλος σε κάθε είδους φορολογικού παραδείσου που επιτρέπει την ομοποίηση χρημάτων, την φοροαποφυγή και την φοροδιαφυγή. Ε, ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you. Ευχαριστούμε την κυρία Σακοράφα. Άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να πάρουν το λόγο. Κύριε much. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να κάνω ένα, ένα σχόλιο ότι ο, το μέγεθος της δημοκρατίας δεν είναι τόσο μεγάλο. Δηλαδή τη δεκαετία του 60 είχαμε τις ελευθέρες ε, ταξιαρχίες, ε, τη Rotter ε, και άλλες Οργανώσει τρομοκρατικέ ε, που δημιουργούσαν ένα κίνδυνο πολύ μεγαλύτερο, σε πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις από ό,τι σήμερα. Ένα δεύτερο σχόλιο. Ε, κύριε Ρενάρτ, δεν σας αντιλαμβάνομαι γιατί μας είπατε ότι η χρηματοδότηση ε, αυτών των ε, ενεργειών, δηλαδή του, του, του World Trade Center, ήταν ουσιαστικά αποτέλεσμα μικροχρηματοδοτήσεων. Ίσως έγινε κάποιο σφάλμα εκεί στην τερμηνία, αλλά πραγματικά δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή η επίθεση που έγινε στο World Trade Center ε, ήταν πάρα πολύ καλά οργανωμένη και χρηματοδοτημένη. Ενώ ε, ε, άλλες επιθέσεις που έγιναν δεν είχαν ούτε καν υποστήριξη από οργανωμένες τρομοκρατικές ομάδες όπως για παράδειγμα το Άζης και χρειάστηκε μόνο ένα λίτρο βενζίνης για να γίνει ότι έγινε. Οπότε ενδεχομένως να υπήρξε κάποιος φορά στη Γερμανία. Πρόεδρος, ε, κύριε θέλετε να σχολιάσετε. Εντάχει, είπα ότι η χρηματοδότηση των διδήμων ήταν μακροοικονομική, μακρο. Ενώ στη Νίκαια και στη Βαρκελόνη ήταν μικροχρηματοδότηση. Ε, η διερμηνία ήταν σωστή, εσείς δεν καταλάβατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Είπα όμως ότι η μικροχρηματοδότηση έχει επικρατήσει. Ως προς τις ερυθρές ταξιαρχίες δεκαετία και 70 χαίρομαι που η Πολωνία δεν είναι στην κατάσταση της Ισπανίας όπου ζούμε καταστάσεις με εκατοντάδες νεκρούς. Δεν το έχετε ζήσει και δεν γνωρίζετε. Το θέμα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο για μας. Και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε την περιπλοκότητα ενός κοινού προβλήματος. Και αυτό που έχει σημασία είναι η κοινή λογική. Οι διάφορες ομάδες λειτουργήσαν κατά τρόπο ώστε να πρέπει να αντιδράσουμε με κοινό τρόπο από το ΕΛΚ μέχρι την ΚΟΕ. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλες τις ομάδες που εργάστηκαν επικοδομητικά για να αντιμετωπίσουμε την κοινή αυτή μάστιγα και επικράτησε η κοινή λογική στη συνεργασία μας. Thank you, Mr. Nart. Ευχαριστούμε τον κύριο Νάρτ. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε στο επόμενο σημείο της σημερινής σας διάταξης, δηλαδή του σημείο 11. συστάσεις προ το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Υπηρεσία εξωτερική δράση σχετικά με τις διαπραγματεύσει για τη Συνολική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωση Αζερβαϊτζάν. Πρώτη λοιπόν συζήτηση αυτού του σχεδίου γνωμοδότησης ε, από τον Σαφρό Νικολάη. Νωρίκα, ε, περιλαμβάνει αυτέ τι συστάσει προ το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Υπηρεσία εξωτερική Έδρασης σε σχέση με αυτή τη συμφωνία. Και η πρακτική τη επιτροπή μα είναι να αναφέρει στου αρμόδιους για την διαπραγμάτευση το τι αναμένει ω προ τα αποτελέσματα τέτοιων συμφωνιών έτσι ώστε η ε, εν λόγω διαδικασία υιοθέτηση αυτή τη συμφωνία να τρέξει ομαλά στο Κοινοβούλιο. Δράτω με τι ευκαιρίε για να υπενθυμίσω στο Συμβουλίο ότι δεν έχουμε λάβει μία σειρά από έγγραφα τα οποία σχετίζονται με αυτές τις διαπραγματεύσεις παρότι δικαιούμαστε νομίμως να τα λάβουμε ως Κοινοβούλιο ε, και ελπίζω να επιληθεί αυτό το ζήτημα το ταχύτερο δυνατό από την πλευρά του Συμβουλίου. Υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος του Συμβουλίου σήμερα εδώ, στην αίθουσα. Ε, εντάξει, αν μας παρακολουθούν τηλεοπτικά να πούμε ότι τους έχουμε αναφέρει το, αυτό το γεγονό επανειλημμένα και το επενθυμίζουμε για μία ακόμα φορά ότι δεν λάβαμε τα σχετικά έγγραφα. Να δώσω το λόγο όμω ε, στην κυρία Νικολάη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Απέστειλα μια επίσημη επιστολή σε εσά και στη Γραμματεία ζητώντα το να, βληθεί η πρώτη συζήτηση αυτών του, του, του σχεδίου γνωμοδότησης και αυτό γιατί γνωρίζω ότι χρειάζεται πολύ σαφεί κατευθυντήρια μέσα από την πλευρά του Συμβούλου στο πλαίσιο αυτών των διαπραγματεύσεων, αφού πρόκειται και για έναν ευαίσθητο τομέα. Δυστυχώ, οι διαπραγματεύσεις ε, τρέχουν, ωστόσο δεν τρέχουν με διαφανή τρόπο, δεν υπάρχει σαφήνεια και δεν γνωρίζουμε το τι ακριβώ συμβαίνει. υπάρχουν τέσσερι δηλαδή διαπραγματευτικοί γύροι σε ό,τι αφορά τον πολιτικό, το πολιτικό τμήμα, έξι σε ό,τι αφορά του ε, ε υπόλοιπου τομεί και δύο γύρου διαπραγμάτευση σε ό,τι αφορά τα εμπορικά ζητήματα. Και βέβαια υπάρχουν διάφορα ε, λεπτά ζητήματα σχέση με αυτή τη διαπραγμάτευση, ειδικότερα σε ό,τι αφορά το σεβασμό ε, του κράτου δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. το Μάιο η ε, επίσκεψή μα επισκέφθηκε, όπω θα θυμόσαστε, το Αζεμπαϊτζάν εκεί στην πρωτεύουσα στο Μπακού ε, και είχε τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με κάποιου αξιωματούχου από εκείνη την πλευρά, ούτω ώστε να γνωρίζει καλύτερα το τι συμβαίνει. Επίση, αναμένω και εγώ αυτά τα έγγραφα από την πλευρά του Συμβουλίου. Σε γενικέ γραμμέ, ε, πράγματι μπορούμε να προβούμε σε κάποιε συστάσει, αλλά δεν θα ήθελα να έχουν τόσο επίσημο χαρακτήρα εν λόγω συστάσεις, ε, γιατί δεν υπάρχει και ένα συγκεκριμένο ε, οριστικοποιημένο χρονοδιάγραμμα σε σχέση με αυτέ τι διαπραγματεύσει και επειδή δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα σε σχέση με αυτέ τι διαπραγματεύσει. Οπότε ε, ζήτησα από την Επιτροπή ε, να και ζήτησα και από σα πρόεδρε να αναβληθεί η παρουσίαση αυτή τη έκταση. Ευχαριστούμε την κυρία Νικολάη. Ζητήσατε λοιπόν να αλλάξει το χρονοδιάγραμμα. Οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων τι έχουν να πούν. Ο κύριος Θα μιλήσω λετωνικά, παρακαλώ. Ε, υποστηρίζουμε την τοποθέτηση της εισηγήτριας. Πιστεύω ότι συντρέχουν οι εξής λόγοι. Τελευταία. Είδαμε πώς πήγε και η επίσκεψη στον Πακού όπου μέλη της Επιτροπής Εκτορικών Υποθέσεων συμμετείχαν. Παρατηρούμε λοιπόν ότι υπάρχει πραγματικά πρόοδος στο Αζερβαϊτζάν. Φαίνεται αυτό, το αισθανόμαστε σαφώς. Πιστεύω λοιπόν ότι φέτος ε, που το Αζερβαϊτζάν θα γιορτάσει και την εκατοστή επέτειό του, από πολιτική άποψη είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διτηρηθεί αυτή η πολιτική ορμή για την πρόοδο Άρα υποστηρίζω την κυρία Νικολάη και την προσέγγιση της. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαμίκινς, λέει ο πρόεδρος, ο κύριος Στατίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το λόγο, πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να πω ευθύ εξ αρχή ότι αντιλαμβάνομαι ότι οι καλέ σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Αζερβαϊτζάν θα ήταν κάτι το αμοιβαία υποφελέ Ωστόσο, δεν πιστεύω ότι είναι η σωστή χρονική στιγμή να προβούμε σε οποιαδήποτε αναβολή τέτοιων εκθέσεων. Οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αζερβαϊτζάν συνεχίζουν ακάτακτες και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προωθεί τις αξίες της. Γιατί σε αυτές βασίζεται και η κατάσταση των δημοσιογράφων και της ε, κοινωνίας των πολιτών στη χώρα αυτή επιδεινώνεται και πάει ο μόνιμος εισηγητής για τις σχέσεις με τη Γεωργία θα πρέπει να αναφέρω τον κύριο Αφκαν Μόχταρλε, την υπόθεση του κυρίου Μόχταρλε, ο οποίος ήταν και ο πρώτος δημοσιογράφος, ο οποίος απήχθη από τη Γεωργία και καταδικάστηκε σε φυλάκιση, εξαετή φυλάκιση στο Αζερμπαϊτζάν. Ανησυχώ, ανησυχώ ιδιαίτερα και θα θέλω να μπει το όνομά του στην έκθεση. Ευχαριστώ με τον κύριο Στατινά. Και τώρα να περάσουμε στην κυρία Φωτίγκα. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και θα ήθελα να υποστηρίξω κι εγώ το αίτημα της εισηγητρίας. Και αυτό για δύο Καταρχάς, συνήθως ε, δείχνουμε μια διακριτική ευχέρεια και μια ευγένεια, αν θέλετε, προς τους εισηγητές και σεβόμαστε την απόψή τους. Φυσικά, όλοι ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερως για τις εξωτερικές υποθέσεις και για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, και έχουμε και τα δικά μας, ε, τις δικές μας ανησυχίες, αλλά νομίζω ότι σε κάποιο σημείο πρέπει να δείξουμε και μια αλφα εμπιστοσύνη προς τον εκάστοτε εισηγητή. Η κυρία Νικολάη είναι ιδιαίτερα έμπειρη ω βουλευτή και γνωρίζω καλά τη δουλειά τη γι' αυτό λοιπόν και τη σέβομαι και την υποστηρίζω. Κατά δεύτερον, η κατάσταση του Αζερμπαϊτζάν ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητη. Ωστόσο έγιναν πολύ θετικέ δηλώσεις και διακηρύξεις από την κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν. Σε ό,τι αφορά και την εκατόστη επέτειο της χώρας. και τα βήματα τα οποία έγιναν για την βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της κατάστασης της κοινωνία των πολιτών. Θεωρώ ότι θα ήταν λογικό και εύλογο να περιμένουμε λίγο και να δούμε κατά πόσο θα υπάρξουν αποτελέσματα, τα οποία και φυσικά εύχομαι να υπάρξουν. Και υπάρχουν και υπάρχει και ένας τρίτος λόγος. Από ιστορικής άποψης, εμείς οι Πολωνοί γιορτάζουμε και την εκατοστή επέτειο της ανάκτησης της ανεξαρτησίας και το Αζερμπαϊτζάν αντιδραμάτισε σημαντικό ρόλο προς την πορεία αυτή για μας. Και γι' αυτό λοιπόν υποστηρίζω το αίτημα αυτό. Thank you, Ms. Ευχαριστούμε την κυρία Φωτίγκα, λέει ο Πρόεδρος. Από την άλλη τώρα, τρεις ομιλητές. Κούτσουκ, Γκριγκούλα και Βάιγκλ. Ποιος θέλει να πάρει πρώτο το λόγο ένα επιχείρημα για να υποστηρίξω την πρόταση της κυρίας Νικολάη. Να σας πω ότι η επόμενη συνάντηση θα είναι στο Μπακού το 2018. Νομίζω ότι είναι καλή ιδέα να δώσουμε στον Πρόεδρο την ευκαιρία να μας παρουσιάσει την έκθεσή του. Και θα ήθελα λοιπόν να ακολουθήσουμε την πρόταση της κυρίας Νικολάη για να γίνει αναβολή της έκθεσης. Μάλιστα, λέει ο πρόεδρος. Κυρία Γκριγκούλα. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Θα μιλήσω λετωνικά και θα αντράξω πραγματικά την ευκαιρία που έχω να μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα. Υποστηρίζω απόλυτα την κυρία Φωτίγκα. Θα πρέπει να, δείξουμε, να δείχνουμε πιο πολύ σεβασμό ενώπιον των εισηγητών. Αυτή η έκθεση δεν έχει φτάσει άλλωστε στη φάση εκείνη όπου θα έπρεπε κάτι να βιαστούμε, να αποφασίσουμε. Δεν υπάρχει λόγος να βιαστούμε. Υποστηρίζω λοιπόν την εισηγήτρια και πιστεύω ότι δικαιολογείται πραγματικά η αναβολή και πολλά ακόμα στοιχεία ενδεχομένω να προσθεθούν στην έκθεση, στην ίδια την έκθεση δεν ναι, ναι. υπάρχει αναφορά και στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί πέρσι περάσαμε διάφορα έγγραφα και έχω να πω ότι συχνά τονίζουμε το ότι έχουν αποφασίσει τα άλλα δεσμικά όργανα και ξεχνάμε τη δική μας τη συνεισφορά. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω την Επιτροπή μας, την Επιτροπή ΑΦΕΤ, να δείξει ίση στάση και σεβασμό για όλες τις ε, δημοκρατίες της περιφέρειας αυτής. Ε, και τονίζω την περίπτωση της Γεωργίας. Και βλέπω ότι, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά το Αζερμπαϊτζάν υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με την Αρμενία. Έχουμε συζητήσει. Αν συζητούσαμε μάλλον την Αρμενία, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα και η στάση μας. Άρα, υποστηρίζω αναβολή. Και πιστεύω ότι τουλάχιστον να περιμένουμε και την αντιπροσωπεία να επιστρέψει. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριο Βάιγκλη τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν νομίζω ότι έχω να προσθέσω κάποιο ιδιαίτερο επιχείρημα σε αυτά που ήδη ακούσαμε. Υποστηρίζω την πρόταση της εισηγήτριας. Αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν διαπραγματεύσει για τη συνεκτική συμφωνία με το Αζερμπαϊτζάν. Ο δρόμο αυτό δεν ήταν ομαλό. Τα τελευταία 1,5-2 έτη είχαμε πολλέ ε, διαφιλονικούμενε απόψει και πολλά καθόδη ζητήματα. Νομίζω ότι σωστά θα κάναμε, καλά θα κάναμε να προετοιμάσουμε σωστά τη διαδικασία αυτή, να λάβουμε υπόψη και όλα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσαμε και ως αντιπροσωπεία της ΑΦΕΤ ε, επισκεφθήκαμε τον Μπακού και το Έρβαν. Νομίζω ότι στο σχέδιο αυτό του κειμένου το θέμα του Ναγκόρνο Καραμπάχ δεν έχει επαρκώς επισήμανθει και αυτό αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα στην περιοχή αυτή. Μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας υπάρχει μια διαρκής πολεμική για το κατά πόσον και πώς θα μπορούσε να επιληφθεί το πρόβλημα αυτό. Νομίζω ότι θα πρέπει να επιδείξουμε ασφαλώς ε, πνεύμα υποστήριξης, αλλά να λάβουμε και παραπάνω πρωτοβουλίες. Τώρα λοιπόν έχουμε την ευκαιρία, έχουμε και το χρόνο, έχουμε και κάποιες ευκαιρίες να ασκήσουμε πίεση στην κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν για τα θέματα ανθρωπινών δικαιωμάτων, τα θέματα τύπου, αλλά ένα-ένα αν θέλετε και να δώσουμε σε κάθε ένα από αυτά το χρόνο που χρειάζεται για να είναι πραγματικά παραγωγικό ο διάλογο με τη χώρα αυτή, γιατί το χρειαζόμαστε τον διάλογο αυτό το παραγωγικό. Και τώρα να ακούσουμε και τον τέταρτο ομιλητή τη Άλντε. Νομίζω ότι πραγματικά είναι ξεκάθαρο το, η θέση σα. ο κ. Αστροβίτσιος. Ευχαριστώ. Δεν είμαστε μεγάλη ομάδα, αλλά σημαντική και με κάθε ευκαιρία εκφράζουμε τις απόψεις μας και επί του θέματος αυτού. Για πολλούς λόγους παίρνω το λόγο. Είπατε ότι δεν υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ Συμβουλίου και Επιτροπής μας και γι' αυτό θα πρέπει να υπενθυμίσουμε το Συμβούλιο για τις υποχρεώσεις του να μας παρέχει σημαντικά έγγραφα, ιδίως όταν πρόκειται για διαπραγματεύσεις. Θα πρέπει να έχουμε τη σωστή πληροφόρηση για να μπορέσουμε να γνωμοδοτήσουμε πριν από οποιαδήποτε ψηφοφορία. Το Αζερβαϊτζάν είναι ένας από τους εταίρους ε, ε, συνεργασίας προς Ανατολάς και είχαμε μία, προβάλλουμε μία συμφωνία για μέσο και μακροχρόνια συνεργασία. Μερικά στοιχεία είναι καλά, άλλα όχι. Στις 12 Ιανουαρίου είδα μία έκθεση όπου έγινε λόγος ε, για την απαγωγή ενός δημοσιογράφου και εκείνος που έκανε την απαγωγή δυστυχώς καταδικάστηκε μόνο σε έξι χρόνια κάθερξη. Αυτό δεν είναι θετικό. Θα ήθελα βεβαίως ε, να συγχαρώ το Αζερμπαϊτζάν για τα ε, εκατοστά γενέθλιά του, αλλά αυτό, αυτή η εκατονταετία ε, έχει ένα αντίτιμο ότι 100 δημοσιογράφοι ή και περισσότεροι βρίσκονται στις φυλακές. Γι' αυτό πολλά θα πρέπει να βελτιωθούν στο κείμενο, χρειαζόμαστε χρόνο και ελπίζω να έχουμε εξισορροπημένες απόψεις και να προωθήσουμε τις σχέσεις μας φυσικά, αλλά υπάρχουν ζητήματα αρχής. Δεν μπορούμε να αποσιωπούμε ζητήματα θεμελιωδών αξιών στο Αζερβαϊτζάν. Γι' αυτό ας ε, λάβουμε μια σωστή, μια έξυπνη απόφαση, έτσι ώστε το κείμενο να αντικατοπτρίζει όλα τα στοιχεία και να λάβουμε και τις πληροφορίες που περιμένουμε από το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λόπες Α, ο κύριος Μέζερης, μάλλον πρώτα ο κύριος Λόπες και μετά ο κύριος Μέζερης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να παρέμβω και να πω για την θέση της ομάδας μας σε σχέση με την έκθεση. Εμείς είμαστε κατά της αναβολής αυτής της έκθεσης. Δεν θεωρούμε ότι θα ήταν ε, σκόπιμο για τις θέσεις μας με το Αζερβαϊτζάν να κάνουμε κάτι τέτοιο και νομίζω ότι η Επιτροπή στο σύνολό της θα πρέπει να λάβει μία απόφαση και ποιες διαδικασίες ακολουθεί. Καταρχήν, ως προς τη διαδικασία θα ήθελα να πω ότι ήρθαμε εδώ, δεν έγινε καμία επίσημη ανακοίνωση για την θέληση αναβολής και ίσα ίσα αναφέρθηκε το αντίθετο πριν, δηλαδή δεν συντρέχουν φυσικά και οι δύο βασικοί λόγοι για την αναβολή. Θεωρούμε ότι ε, αν αναβάλουμε δεν θα έχουμε μία εργαλειοθήκη για να μπορέσουμε να επηρεάσουμε μία ενδεχόμενη απόφαση. Γι' αυτό όχι μόνο αναβάλουμε, αλλά ε, αυτό περιοριζόμαστε μη διαθέτοντας ένα μέσο πίεσης. Και τρίτον, όχι μόνο περιορίζουμε ένα μέσο ή μία εργαλειοθήκη που έχουμε στα χέρια μας, αλλά στο τέλος με την αναβολή δεν θα φτάσουμε σε μία συμφωνία και δεν θα μπορέσουμε να πιέσουμε. Και δεν νομίζω ότι θα ανακύψουν νέα γεγονότα που θα μας οδηγήσουν σε μία αλλαγή θέσης. Γιατί δεν πρόκειται να αλλάξουν ουσιαστικά δεδομένα για αυτή την αναβολή. Δηλαδή, αν ανέκυπτε κάτι νέο, τότε πραγματικά να γινόταν αναβολή. Αλλά δεν έχει πια ε, προκύψει ένα τόσο ε, ουσιαστικό γεγονός που να μας οδηγεί σε κάτι τέτοιο. Καταλαβαίνω ότι οι σχέσεις μας είναι πιεσμένες τα τελευταία χρόνια. Θα πρέπει να προβάλλουμε μία δική μας στρατηγική για να επιβάλλουμε ε, τη θέση μας. Ξέρουμε τις ε, περιφερειακές ε, σειράξεις, τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά δεν άλλαξαν τα πράγματα τους τελευταίους μήνες για να μπορέσουμε να πούμε ότι «Α, αυτό το γεγονός ε, αποτελεί μια πραγματική τροχοπέδη. Το χειρότερο είναι να μην υπάρχει έκθεση. Δεν έχει νόημα να αυτοπεριοριζόμαστε χωρίς κανένα αντίκτυπο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Λόπες. Τώρα, ο κύριος Μέζεριτς έχει το λόγο και μετά ο κύριος Σνάρτ. Ε, ευχαριστώ. Ως ε, σκιώδης, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για ένα κείμενο που θεωρούμε ότι είναι πολύ καλό σημείο εκκίνησης και θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια πολύ καλή έκθεση ως προς το διαδικαστικό. Δεν πρόκειται για μια κοινοβουλευτική διαδικασία, πρόκειται και για ε, θέμα διεθνούς πολιτικής. Γι' αυτό υπάρχει κάποιος λόγους για αναβολή ψηφοφορίας μετά από τις διαπαραματεύσεις με την αντιπροσωπεία στο Μπακού. Πιστεύουμε όμως ότι το να γίνει μία συζήτηση πριν από τις διαπραγματεύσεις, τότε θα ενισχύσουμε τη θέση των διαπραγματευτών στο Μπακού. Δηλαδή, θα πρέπει να ορίσουμε τις προσδοκίες μας και μόνο αν έχουν αλλάξει τότε θα αναβάλουμε. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε ποιες είναι οι προσδοκίες μας καταρχήν. Γι' αυτό θα ήταν σκόπιμο να γίνει μια συζήτηση πριν μεταβεί η αντιπροσωπεία στο Μπακού και ενδεχομένως να αναβάλουμε την ψηφοφορία και μόνο. Γνωρίζουμε τις σειράξεις στην περιοχή εκείνη της Ευρασίας, αλλά δεν νομίζουμε ότι θα επιληθούν με αυτόν τον τρόπο. Είναι προαιώνιες οι σειράξεις Απλώς θα πρέπει να προβάλλουμε υποδείξεις για να βελτιώσουμε το πλαίσιο διαπραγματεύσεων. Σας ευχαριστώ πολύ ο κύριος Νάρτ. Το, στο Αζερβαϊτζάν το πρόβλημα ε, υπάρχει εσωτερικό και εξωτερικό πρόβλημα. Υπάρχει ε, ανελευθερία τύπου και συνεταιρίζεστε και ως προς το εξωτερικό έχουμε να κάνουμε με τον Αγκόρνο ε, Καραμπάχ. Το ίδιο ισχύει και στη Λιβύη με μια κυβέρνηση ανδρίκελο την οποία δεν αναγνωρίζει κανένας. Το ίδιο ισχύει και στην Παλαιστίνη με το πρόγραμμα ειρήνης των ΙΠΑ και του Νετανιάχου και στην Ιεμένη όπου αναγνωρίστηκε μία κυβέρνηση μαριονέτα. Αυτά συμβαίνουν παντού. Και εδώ μιλάμε για τις συμφωνίες της Μαδρίτης και του Μίνσκ που αποτελούν λύση του προβλήματος. Όταν απελευθερώθηκε ε, ε, το Αζερβαϊτζάν και η Γεωργία, τότε στην Οσετία και στο Ναγκόρνο Καραμπάχ δεν δέχτηκαν να προσχωρήσουν σε αυτές τις δύο δημοκρατίες. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να ε, λέμε ότι πρόκειται για θέμα αυτοδιαχείρισης και αυτοδιάθεσης. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα, διότι έτσι θα δημιουργήσουμε δύο ή τρία μέτωπα. Γιατί η λύση του Ναγκόρνο Καραμπάχ δεν μπορεί να είναι η ίδια λύση για την Οσετία ή για την ε, Κρυμαία. Γιατί η πίεση των Αρμενίων οδήγησε σε ένα προηγούμενο και έτσι η Ρωσία το χρησιμοποίησε για την Κρυμαία. Δηλαδή η Αρμενία έχει μία μεγάλη στρατιωτική βάση στον Κάφκασο. Εάν λοιπόν εθελοτυφλούμε και δεν κατανοούμε το φαινόμενο του Ναγκόρνο Καραμπάχ, της Οσετίας και της Κρυμαίας δείχνει ότι είμαστε αντιφατικοί και προς τις δύο ή τρεις κατευθύνσεις. Σας ευχαριστώ. Νομίζω πως ακούστηκαν όλα τα επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές, υπέρ και κατά δηλαδή, τις ε, αναβολές. Ε, διαφορετικέ απόψει ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα. Πάντως ε, θεωρώ πως όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι δεν θα γίνει σήμερα η πρώτη εξέταση του σχεδίου της έκθεσης. Αυτό είναι προφανές. Τώρα, ε, Άλντε και η συγκήτρια μας ζήτησαν να αναβάλουμε την έκθεση ο κύριος ε, Μίτερς ήταν υπέρ. Ε, ναι, ο κύριος ε, Λόπες εκ μέρους της πολιτικής ομάδας κατά, το ΕΛΚ είναι κατά και η πράσινη επίσης όπως εκφράσαμε ο κύριο Μέζερης είναι κατά. Και για το ECR, α, με τη σειρά του, α, είναι υπέρ. Οπότε, θα ήθελα στο πλαίσιο του διευρυμένου Πρέπει να συζητηθεί αυτό με τους εκπροσώπους δηλαδή του, των πολιτικών ομάδων γιατί θα πρέπει νομίζω να λάβουμε υπόψη μας ε, πολλά από τα επιχείρηματα που εξέθεσαν και οι δύο πλευρές. ειδικότερα ως προς ε, την ισότιμη μεταχείριση της οποίας θα πρέπει να την χάνουν όλοι οι συγητές και όλες οι εκθέσεις. ας λοιπόν προσπαθήσουμε εκεί στο Διευρυμένο Προεδρείο να φτάσουμε σε μια συμφωνία. α μην ε, διαφωνήσουμε σήμερα εδώ. Πότε θα λάβει η χώρα επόμενη συνεδρίαση. «25 Φεβρουαρίου είναι η επόμενη συνεδρίαση, αλλά μπορούμε να κάνουμε και μια γραπτή διαδικασία. Γιατί πραγματικά ακούστηκαν κάποια πολύ εύστοχα επιχειρήματα από την πλευρά των συναδέλφων. Ε, πάντως ε, το Έλκ και οι σοσιαλιστέ, μάλλον η πλειοψηφία δηλαδή, είναι κατά τη αναβολή. Αλλά θα δούμε, θα το συζητήσουμε λοιπόν στο Δημοτικό Προεδρείο. Η κυρία Νικολά έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για αυτό το συμπέρασμα. Ε, θα ήθελα να είμαι λίγο πιο συγκεκριμένη. Δεν αξίωσα την αναβολή τη έκθεση. Ζήτησα την αλλαγή του χρονοδιαγράμματος. Έχουμε να κάνουμε μια έκθεση που αφορά σε συστάσεις προς το Συμβούλιο. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και πιο σοβαροί. Αλλά από εκεί και μετά δεν θα πρέπει να είμαστε πιο επίσημες ως αυτές τις συστάσεις, γιατί η κατάσταση είναι πολύ ευαίσθητη, πολύ λεπτή. Άρα λοιπόν, το ζήτημα είναι ένα ζήτημα αξιοπιστία. Θέλουμε να ασκήσουμε απλώ και μόνο κριτική στο Αζερμπαϊτζάν. Ναι, μπορούμε να το κάνουμε, μπορούμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Αλλά παραμένουν κάποια άτομα που παραμένουν κρατούμενοι Και γι' αυτό θα ήθελα να υπάρξει μια σαφή τοποθέτηση και από την πλευρά του Αζερβαϊτζάν σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση μπορούμε να περιγράψουμε πάρα πολύ γλαφυρά τα όσα συμβαίνουν εκεί, χωρί όμω να επιτύχουμε τίποτα παραπάνω. Και κάτι τέτοιο υπονομεύει τη θέση μα και υπονομεύει την αξιοπιστία μα. Εάν θέλουμε να έχουμε λοιπόν μια εταιρική σχέση με το Αζερβαϊτζάν, θα πρέπει ακριβώ να δράσουμε ω εταίρο. Δεν έχω δηλαδή εγώ κάποια, κάποιο άλλο στόχο, αλλά λέω για να είμαστε αξιόπιστοι ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως Ευρωπαίοι πολιτικοί, θα πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι σε, σε σχέση με αυτές τις συστάσεις που θα κάνουμε. Μετά, ένα δεύτερο ζήτημα που αναφέρθηκε από τον συνάδελφό μου είναι το ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σαφής και συνεχιζόμενη συνεργασία με το Συμβούλιο, πράγμα το οποίο δυστυχώς δεν ισχύει στην περίπτωση αυτή, δηλαδή των διαπραγματεύσεων με το Αζερμπαϊτζάν. Ε, και ελπίζω πω οι συστάσεις μα θα αποτελέσουν μια συνεισφορά προς τις διαπραγματεύσεις. Ε, όμως όμω είναι πιο επίσημε αυτέ οι συστάσει, λάβουν ένα πιο επίσημο χαρακτήρα, τότε ουσιαστικά θα εξυπηρετήσουν μόνο τα πιο σημαντικά ζητήματα, δηλαδή τα οικονομική φύση ε, ζητήματα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που ελπίζω να έχουμε και στο οποίο να καταλήξουμε είναι μια καλή έκθεση η οποία τελικά, ε, τις οποίες οι συστάσεις θα μπορούσαν να πραγματικά αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Ευχαριστώ, λέω ο πρόεδρος ε, την κυρία Νικολάη. Ε, και με ενδιαφέρον άκουσα αυτό που είπατε, ότι ζητήσατε απλώς μια μεταβολή του χρονοδιαγράμματος και όχι αναβολή της έκθεσης, που για μένα είναι αρκετά παρόμοιο. Αλλά ας δώσω τώρα το λόγο στον επικεφαλής της διαπραγματευτικής σας ομάδας, τον κύριο Λουκ Ντεβίνιεν. Θέλετε να πείτε δύο λόγια ή τι προτείνετε εσείς ε, θα πρέπει να αλλάξει το χρονοδιάγραμμα ή όχι. Παρακαλώ κύριε Ντεβίνια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και καλημέρα σε όλα τα αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι δύσκολο εγώ να τοποθετηθώ βέβαια σε ό,τι αφορά την απόφαση που θα λάβετε, αλλά μπορώ να σε ενημερώσω σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις που έχουν, έχουν τρέξει μέχρι τώρα και βέβαια είμαστε στι διάθεσή να σας ενημερώσουμε και στο μέλλον σε σχέση με αυτές τις διαπραγματεύσεις. Πάντως ε, προφανώς δεν ε, είναι δική μου δουλειά εγώ να σχολιάσω <laughs> και να τοποθετηθώ σε ό,τι αφορά αυτή την πρόταση που έγινε για μεταβολή του χρόνου διαγράμματο. Ε, ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Κρίμα που δεν μπορείτε να τοποθετηθείτε. Ε, εν ακούστηκαν όλα τα επιχειρήματα, όλα τα υπέρ και όλα τα κατά και θα συζητηθεί το ζήτημα περαιτέρω στο διευρυμένο πρόεδρο. Σα ευχαριστώ λοιπόν όλου όσου συμμετείχατε σε αυτή τη συζήτηση. Και τώρα Ε, περνάμε στο επόμενο σημείο της μέσης διάταξης, αλλά έχουμε ολοκληρώσει μισή ώρα νωρίτερα. Οπότε διερωτώ υπάρχει ήδη από τώρα κάποιος εκπρόσωπος από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για να συζητήσουμε το σημείο σε ό,τι αφορά τους Ροχίνγκια. Um, the External Action Service will be with us in 10 minutes. Η υπηρεσία εξωτερική δράσεως θα έρθει σε 10 λεπτά. Ξεκινήσουμε, συνεχίζουμε λοιπόν την συνεδρίαση στις 11 παρα 20. Right, dear colleagues, we can continue our meeting. It's... Συνάδελφοι, να ξαναξεκινήσουμε. Έχει πάει και 11 παρατάρτο. Item number 12. Στο 12 λοιπόν της ημερήσιας διάταξης. Θα κάνουμε ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για την κατάσταση των Ροχίνγκα στη Μιαμάρ. Και θα ήθελα να σας επενθυμίσω ότι η Επιτροπή ΑΦΕΤ ε, της και να συμμετέχει στην αποστολή στο Μιανμάρ για τις 12 ε, έως 16 Φεβρουαρίου. Και οι αυτόπτες μάρτυρες μας ε, περιγράφουν την κατάσταση στο Ροχίνγκα ως απελπιστική από τότε που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2017 η επίθεση στο Ροχίνγκα από τους ε, ανάρτες και πρέπει να σας πούμε ότι η πρόσβαση στις ανθρωπιστικές οργανώσεις είναι πιο δύσκολη, όλο και πιο δύσκολη και έχουν γίνει κοινώσεις πολλών. Σύμφωνα με τον υπηρεσία του ΟΗΕ, πάνω από 600.000 άτομα έχουν μεταβεί, έχουν φύγει στον Μιαμάρ από πέρσι και ζουν πλέον σε κατασκηνώσεις, σε... Να σας πω ότι α, Επιπλέον η Μιανμάρ αποτρέπει όλες τις παροχές βοήθειας από τις ε, περιοχές στην Βόρειο κράτος του Ρακίνε. Και έχουμε μαζί μας λοιπόν τους εκπροσώπους της ε, ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης σήμερα, ο κύριος David Haley, Daly, ο οποίος είναι επικεφαλής του τμήματος για την Νοτιοανατολική Ασία και την κυρία Ισαμπελ Τελάτρε, η οποία είναι επικεφαλής του τμήματος περιφερειακών σχέσεων με την Ανατολική Ασία οι οποίοι έχουν έρθει εδώ μαζί μα για να μα παρουσιάσουν τι πρόσφατε εξελίξει και τι προσπάθειε τη διεθνού κοινότητα και τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να αλλάξει η στάση τη ε, κυβέρνηση του Μιανμάρα. Να δώσουμε λοιπόν πρώτα το λόγο στον κύριο Ντέιλι και μετά στην κυρία Ντελάτρ. Να σας υπενθυμίσω ότι το επόμενο θέμα θα ξεκινήσει στις 11.30 όταν θα έρθουν και οι προσκεκλημένοι από το Ιράν. Ο κύριος Ντέιλι έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και όντω ε, τιμή και χαρά που βρίσκομαι εδώ στην Επιτροπή σα του Κοινοβουλίου, την Επιτροπή Εκτρικών Υποθέσεων. Κάποια γενικά σημεία, επιτρέψτε μου, καταρχά. Ε, όπως ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ε, πολιτικά σε επαγρύπνηση μέσω εκτενούς ανθρωπιστικής αρρωγής για να βοηθήσει με τον καλύτερο τρόπο την, τρόπο, την κρίση των προσφύγων των Ροχίνγκα. Και έχουμε σημαντική πολιτική και οικονομική παροχή βοήθειας προς τον Μπαγκλαντές και τη Μιαμάρ. Η πολιτική υποστήριξη μεταξύ άλλων γίνεται σαφής με την προσωπική συμμετοχή και δέσμευση της ε, είπα της εκπροσώπους η οποία έχει επισκεφτεί α, ε, καταβλισμούς προσφύγων, έχει συναντηθεί με τους πολιτικούς ευθύνοντες και έγινε και μία συνάντηση στο Ρακάι με τα το Νοέμβριο στα πλαίσια τη συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικό. Και καλωσορίζουμε λοιπόν το γεγονό ότι το Κοινοβούλιο και η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου σύντομα θα επισκεφτεί και την Μιαμάρ και τον Μπαγκλαντέ και τους καταβλισμούς των προσφύγων στο Κοξής Μπιζάρ. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για να είναι οι εθελοντικές επιστροφές αξιοπρεπείς και να βασίζονται σε μια αμοιβαία συμφωνία και να προαγάγουμε και να λύσουμε τις βασικές αιτίες. Να πω δύο λόγια για τη συμφωνία επαναπατρισμού, η υπογραφή μεταξύ Μπαγκλαντές και Μιανμάρ για την επιστροφή των ατόμων αυτό από το Ρακάν ήταν ένα σημαντικό πρώτο βήμα για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, η οποία τελικά θα καταλήξει στην επιστροφή των ατόμων αυτών. Η εφαρμογή λοιπόν τη διευθέτηση αυτή θα πρέπει να παρακολουθηθεί προσεκτικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό τη, για να εξασφαλίσουμε ότι συνάδει πλήρω με το διεθνέ δίκαιο. Ο ρόλο του ΟΗΕ, πιστεύουμε, και κυρίω ε, του, της είπατε του είπατε εκπροσώπου για την, τα άτομα που τα προσφυγικό ζήτημα είναι σημαντικό. Και ο λόγος λοιπόν που μάλλον η συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών θα ελεγχθεί επίσης, γιατί φοβόμαστε ότι ενδεχομένω να μην υπάρχει συμμετοχή όλων των φορέων στην εφαρμογή και αμφιβάλλουμε για το κατά πόσον τηρούνται τα, τα διεθνή πρότυπα για την επιστροφή, την αξιοπρεπή επιστροφή των ατόμων αυτών. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να παρακολουθούμε τις δύο χώρε, στα πλαίσια και του ΟΗΕ. Από πλευρά της Μιανμάρ, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει την ισορροπημένη της πολιτική που αποτελείται από πολιτική πίεση στα σκόλπου στο ΟΗΕ, στο Συμβούλιο Ασφαλείας, στη Γενική Συνέλευση, στο, στη συνέλευση, στο Συμβούλιο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και την επικοδομητική, ε, επικοδομητικές επαφές με τη Μιανμάρ. Από πλευρά του ΟΗΕ η διερευνητική αποστολή στην Μιανμάρ η οποία ζητήθηκε πέρσι εξάντλησε την εντολή της, η οποία ολοκληρώθηκε το φθινόπωρο και ακολούθησε και ένα ψήφισμα από το OIC και άλλο ένα ψήφισμα στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 5 Δεκεμβρίου. Υποστηρίχθηκε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση το ψήφισμα αυτό. Σε ό,τι αφορά τη λογοδοσία τα ανθρώπινα δικαιώματα, σημειώσαμε τις διάφορες ε, καταγγελίες και μαρτυρίες ε, μικείο του ΟΗΕ διευρυντικών αποστολών για τις σοβαρές συστηματικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εν ώψη όλων αυτών η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι είναι λυπηρό το γεγονός ότι η Μιαμάρ δεν έκανε σοβαρές έρευνες ε, μέχρι σήμερα. Κατά δεύτερον, δεν συνεργάζεται ακόμα με την ερευνητική αποστολή διερευνητικές αποστολές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και κατά τρίτον πρόσφατα σταμάτησε τη συνεργασία με τον ειδικό, την ειδική απεσταλμένη και εισηγήτρια του ΟΗΕ, η κυρία Λί. Καλώς ορίζουμε τη γενικότερη δέσμευση της κυβέρνησης να εφαρμόσει τις συστάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής για το ΡΑΚΑΙΜ, η έκθεση ΑΝΑΝ όπως αποκαλείται. Και καλώ ορίζουμε επίση τι πρόσφατες ανακοινώσει και δηλώσει που έγιναν σε ό,τι αφορά το στόχο για την ε, αφαίρεση κάποιων καταβλισμών Ροχίνγκα στην κεντρικό Ρακάιμ. Αλλά πιστεύουμε ότι θα πρέπει να καταρριστεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράση από την κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την έκθεση Ανάνς με θεματικέ και γεωγραφικέ προτεραιότητε. Αυτό θα βοηθήσει την κινητοποίηση, πραγματική κινητοποίηση διεθνού και ευρωπαϊκή υποστήριξη. Η βελτίωση λοιπόν των συνθήκων ε, διαβίωσης στην, ε, στο ΡΑΚΑΕΜ θα βοηθήσουν και θα δημιουργήσουν ένα ευρωικότερο κλίμα σε ό,τι αφορά την εθελούσια, την εθελοντική επιστροφή όσων έχουν διαφύγει στον Μπαγκλαντές. Σε ό,τι αφορά την αρρωγή, στην διάσκεψη στη Γενέβη τον Οκτώβριο, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποσχέθηκε την πιο υψηλή ε, αρρωγή σε σχέση με τους υπόλοιπους δουλειτές. 30 εκατομμύρια φρέσκο χρήμα με 170 εκατομμύρια δολάρια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της ουσιαστικά δίνουν τη μισή από τη συνολική βοήθεια από αυτή που έχει υποσχεθεί να χορηγηθεί. Τα επιπρόσθετα λοιπόν 30 εκατομμύρια για τις ανθρωπιστικές ανάγκες των Ροχίγκα στο Μπαγκλαντές και για τις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων που τους υποδέχονται. Από τα χρήματα αυτά λοιπόν η ανθρωπιστική βοήθεια θα θέλει 10 εκατομμύρια, τα οποία έχουμε ήδη δεσμευτεί να δώσουμε, και 5 εκατομμύρια ε, δολάρια για την καταχώρηση των προσφύγων. Αυτό ήδη έχουμε υποσχεθεί ότι θα το χορηγήσουμε στις αρχές του μήνα. Και είμαστε λοιπόν στο, στα 78 εκατομμύρια για τους Ροχίνγκα από τις ε, Φρέσκες αυτές οι υποσχέσεις λοιπόν των 20 εκατομμυρίων, 15 εκατομμυρία θα έχουν σκοπό χρηματοδότηση μέσω πρόθεσμων και μακροπρόθεσμων λύσεων. Και μία αποστολή για την αξιολόγηση των αναγκών έχει λάβει χώρα ήδη για να εντοπιστούν ενδεχόμενα σχέδια τα οποία θα χρειάζεται να υλοποιηθούν από πλευρά τη Μιανμάρ τώρα. Είναι φιλόδοξη η ατζέντα για τα μέτρα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποστηρίξει ένα σημαντικό πρόγραμμα καταρχάς για τη μεταρρύθμιση του τομέα της εκπαίδευσης για ύψους πάνω από 120 εκατομμυρίων ευρώ. Και αυτό συνάδει με τις συστάσεις της έκθεσης ΕΝΑΝ. Πρόεδρε, στο σημείο αυτό ολοκληρώνω τα εισαγωγικά μου σχόλια και με χαρά να απαντήσω ό,τι ερωτήσει ενδεχομένως έχουν να μου απευθύνουν οι ευρωβουλευτές να δώσω το λόγο ενδεχομένω στη συνάδελφο, μήπω θέλει να πάρει το λόγο να μιλήσει για τον Μπαγκλαντέ. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν έχω να προσθέσω πολλά από τη δική μου πλευρά. Απλώς ε, σε σχέση με αυτή την ε, αποστολή αποτίμησης θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα για να βοηθήσουμε το Μπαγκλαντές να αντιμετωπίσει αυτή την ροή προσφύγων τους τελευταίους μήνες και ε, παρά αυτή την συμφωνία μεταξύ Μπαγκλαντές και Μιανμάρ για την επιστροφή των Ροχίνγκια θα ε, μάλλον αναμένουμε να παραμείνουν στο Μπαγκλαντές για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό χρειάζεται βοήθεια όχι μόνο ανθρωπιστικής φύσης, αλλά ε, θα πρέπει να συνδεθεί και με αναπτυξιακή βοήθεια γνωρίζοντας ότι αυτή η ροή προσφύγων έχει μεγάλη επίπτωση στις υποδομές ε, και κοινότητες υποδοχής που μιλούν για επιδίνωση του περιβάλλοντος και ούτω καθεξής. Υπάρχουν λοιπόν επιπτώσεις στο Μπαγκλαντές και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να βελτιωθεί η κατάσταση ως προς την φυσική κατάσταση και αντιμετώπιση, θα πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί αυτό το πλαίσιο, γιατί αρχικά είχαν συμφωνήσει οι δύο χώρες να αρχίσει η ροή σήμερα. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αρχίσει ο επαναπατρισμός σήμερα, αλλά όπως είπε και ο συνάδελφος, για μας το πρόβλημα είναι η ύπατη αρμοστία να είναι αυτή που να εξασφαλίσει την εθελούσια και αξιοπρεπή επιστροφή των προσφύγων ο υπεύθυνο από τη δική μου ε, υπηρεσία ε, όρισε ακριβώς αυτό το πλαίσιο ότι θα υπάρξει συνεργασία και του Υπουργείου Εξωτερικών έτσι ώστε από πλευράς ε, Μπαγκλαντές να υπάρχει συνεργασία με την ύπατη αρμοστία για τους πρόσφυγες. Δεν προβλέπεται κάτι από πλευράς Μιανμάρ, αλλά τουλάχιστον οι οικογένειες και ε, οι γυναίκες να μπορέσουν να συνενοηθούν με την οικογένειά τους και η ύπατη αρμοστία θα είναι παρούσα έτσι ώστε να είναι Η πρώτη συνάδελφος έχει το λόγο, βρεθεί εδώ σήμερα και ζητά συγνώμη για την απουσία της μαζί με την Νίνα και άλλους συναδέλφους εξωτερικών μας εκπλήσει γιατί το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών δεν έχει φτάσει σε συμπεράσματα από τον Οκτώβριο παρά το γεγονός ότι γίνονται αυτοί οι εκτοπισμοί που έχουν λάβει χαρακτήρα γενοκτονίας και δυστυχώς και χτεν επεκτείνονται οι κυρώσεις κατά εκείνων που είναι υπεύθυνοι για τη βία ιδιαίτερα των στρατιωτικών. Η Συμφωνία Επαναπατρισμού επίσης έχει καθυστερήσει, αλλά όταν αρχίσει η εφαρμογή, πώς είμαστε σίγουροι ότι δεν θα... Μετά από τις ε, δηλώσεις σας, μπορείτε να μας εξασφαλίσετε ότι ότι ε, οι αρχές του Μιανμάρ δεν θα παραβιάσουν τα δικαιώματα των Ροχίνγκιας που επαναπατρίζονται, διότι όσοι βρίσκονται σε αντιμετωπίσουμε την κατάσταση όπου οι πρόσφυγες δεν θα έχουν δικαίωμα στέγασης μετά τον επαναπατρισμό ή καθυστερώντας την εκπαίδευση των παιδιών των Ροχίνια. Και πέμπτον, πώς θα βρούμε μακροχρόνιες λύσεις για τους ε, Ροχίνια που δεν θέλουν να επιστρέψουν λαμβάνοντας υπόπανου και της γεωργίας έτσι ώστε οι μεταρρυθμίσεις να οδηγήσουν στην αυτάρκεια των προσφύγων και τέλος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πώς μπορεί να συνδράμει τις ε, ε, δικές σας δράσεις ιδιαίτερα μετά την Είστε σήμερα εδώ μαζί μας το πρωί. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μούντι. Ο κύριος Ναρτούρα για Αυτό που, που έχουν οι βουδιστές στην δυτική κουλτούρα φαίνεται ότι ένας βουδιστής μπορεί να είναι και που έχουν οι βουδιστές στην δυτική κουλτούρα φαίνεται ότι ένας βουδιστής μπορεί να είναι και όπου ε, ζει αυτή η εθνότητα. Όλοι οι πόλεμοι μετά το 47 στο τη συμβίωση της ε, Βυρμανίας έτσι ώστε να είναι η Βιρμανία των Βιρμανών με, με ένα πρόβλημα όχι ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά εθνοτικού και εθνικού προσδιορισμού όπου αποκλείονται δυστυχώς οι Ροχίνγκια θα βρίσκονται για πολλά χρόνια το Μιανμάρ που έχει την ίδια προσέγγιση με τους Χαν. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση πέρα από τη Σκνία, η Μαλαισία, η Ινδονησία και το ε, Μπαγκλαντές που βρίσκονται κοντά δείχνει ότι έχουμε την κατάσταση και όχι μόνο θεωρητικά αλλά έμπρακτα με οικονομικό αποκλεισμό. Thank you, And... Ευχαριστούμε τον Χαβιενάρτ. Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε, και ευχαριστώ τους δύο μελετές για τις δηλώσεις που έκαναν. Εγώ θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα. Εμείς υποστηρίζουμε λοιπόν την έκθεση Κοφεανάν ε, για την ανοικοδόμηση ε, της περιοχής Ετουράκ για να υπάρξει καλύτερη συνεργασία. Η έκθεση Ανάν δεν αναφέρεται όμως στα ζητήματα της παραβίασης των ανθρωπίνων ανοικοδόμηση ε, της περιοχής Ετουράκ για να υπάρξει καλύτερη συνεργασία. Η έκθεση Ανάν δεν αναφέρεται όμως στα ζητήματα της παραβίασης των ανθρώπων κυβέρνηση Δηλαδή μια αποστολή η οποία καλείται να διαρευνήσει αυτές τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η οποία τελικά όμως δεν μπορεί να φέρει πέρα σε αυτή την αποστολή. Ε, και ταυτόχρονα η κυβέρνηση και η ε, Σουρκή λέει ότι ε, δεν πρέπει να, κάνουμε να κάνουμε είναι να ασκήσουμε πιέσεις και να πούμε ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί να θεωρεί η κυβέρνηση της Μέρμαρ και η πως όλες αυτές οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα περάσουν έτσι, χωρίς να υπάρξουν κυρώσεις. Πλαίσιο, να εξετάσουμε δηλαδή πιο προσεκτικά τα όσα αφορούν την ατιμορρησία εδώ. Θα πρέπει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει μια πιο σαφή στάση απέναντι σαν ε, Δηλαδή όταν εκείνη λέει ότι θέλει να διερευνήσει αυτές τις ε, ε και θέλει να οδηγήσει τους υπευθύνους ενώπιον της δικαιοσύνης, Βέβαια ε, με την ε, επίσκεψη που θα λάβει η χώρα του σοσιαλιστές. Ε, σας ευχαριστώ πολύ που με δέχεστε εδώ. Είμαι εκπρόσωπος των χωρών ΑΣΕΑΝ. Έχω δύο ερωτήσεις να... Σε περίπτωση που ε, δεν θα υπάρξει καταδίκη των αυτούργων αυτών των εκδιώξεων μεταξύ ιδιαίτερα των στρατιωτικών, ε, τι προβλέπετε να γίνει. Τώρα, ως προς τις οικονομικές ε, επιπτώσεις, η εξωτερική ότι δεν τηρούνται πια οι προϋποθέσεις η συμφωνία. Ευχαριστούμε τον Μαρκ Καραμπέλα. Και έχω έναν ακόμα. Μερθεί τον κύριο Μπετίνε τώρα. Ευχαριστώ. Προσία συμφωνώ με αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Θα ήθελα να ασχοληθώ με ένα πολιτικό ζήτημα προοπτικής. Εμείς όταν κέρδισε η Σαν την ε, προεδρία της χώρας, η Γερμανία, ε, αφορούσε την αντιμετώπιση, ίση αντιμετώπιση των εθνοτήτων και εθνοτικών μειονοτήτων σε σχέση με τη στρατιωτική χούντα που είχε αντιμετωπίσει τις εθνότητες μέσα σε ένα κύμα βίας, σιώπησε. Και προέβαλε ορισμένες εθνικιστικές κορώνες σε σχέση με το βιρμανικό κράτος. Ήδη τότε είχαμε... Μίλησα για αυτά τα ανοιχτά ζητήματα. Άρα το θέμα δεν αφορά μόνο τους Ροχίνια, αν και εδώ πρόκειται για ένα σκανδαλώδες ζήτημα, πρόκειται για τους Σαν Κατσίν, Καρίγιαν, όλες αυτές τις εθνότητες, ιδιαίτερα τους Σαν. Και νομίζω ότι δέκα χρόνια μετά θα έπρεπε να γίνει ε, μία ε, δημοσκόπηση και ένα δημοψήφισμα για αυτές τις εθνότητες ε, στο βορρά της χώρας, στη Γερμανική θα πρέπει να κατανοήσουμε πέρα από την επίγουσα κατάσταση τι σκέφτεται η πρόεδρος της ε, Βυρμανίας, η κυρία Σανσουσί, σε σχέση με αυτές τις τάσεις αυτονόμησης αυτών των εθνοτήτων. Αυτό των ε, εθνοτήτων. Αυτό θα πρέπει να το δούμε και στα πλαίσια της αντιπροσωπείας μας, ε, στη μετάβασή μας δηλαδή ως άφετ στη Βυρμανία. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μπετίνη. Δεν υπάρχουν άλλα σχόλια λοιπόν από πλευρά σα. Ποιο θέλει να ξεκινήσει, παρακαλώ, κύριε Τέιλι, φαντάζομαι να ξεκινήσετε εσεί. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρα, να ευχαριστήσω και του βουλευτέ ε, για τα ζητήματα που έθεσαν και για τι ερωτήσει του. Ιδιαίτερα ή κάτι όμως περισσότερο. Τις δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίω ε, του Συμβουλίου ε, Εξωτερικών Υποθέσεων. Προφανώ. το θέμα αυτό απασχολεί ιδιαίτερα το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και πριν από κάθε Συμβούλιο στο πλαίσιο αυτού και για την απόφαση αυτή. Με την απόφαση αυτή, μάλλον σχετίζονται πολλά από τα θέματα που έθεσαν οι Ευρωβουλευτέ σε ό,τι αφορά δηλαδή το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ό,τι αφορά τι στοχευμένε κυρώσει κατά συγκεκριμένων προσώπων σε ό,τι αφορά το ήδη φυστάμενο όπλων και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα ζητήματα αποτελούν τμήμα των διαβουλεύσεων στα πλαίσια του Συμβουλίου Εκτορικών Υποθέσεων της ε, βαθιάς ρίζας των προβλημάτων αυτών. Η ιστορία προφανώς ε, διδρα... Νομίζω ότι θα πρέπει να τα έχουμε πάντα υπόψη μας σε ό,τι αφορά και τις προσδοκίες μας ασφαλώς. Ασφαλώς ε, και θα προτιμούσαμε μια κατάσταση στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε απλά να αναστρέψει τις ε, ισορροπίες ασκώντας πίεση στην κυβέρνηση του Μιαμάρ και άλλες κυβερνήσεις. Αλλά ασφαλώς έχουμε υπόψη μας τις δυσκολίες. Παρόλα αυτά, συνεχίζουμε να τονίζουμε τα σημαντικά να υπάρξει μια κατάσταση όπου οι πρόσφυγες θα μπορέσουν και θα μπορούν να επιστοχείς και τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεθνούς κοινότητας. Θα πρέπει να φροντίσουμε να είναι εθελούσια η επιστροφή και η επιστροφή τελικά να τα ε, υγειονομικά, υγειονομικές Και αυτό με τη σειρά του φυσικά προκαλεί άλλα τεράστια προβλήματα. Αμα επιστροφών και τι έκταση θα είναι. Αυτά όλα θα πρέπει να τα δούμε με στενή συνεργασία με τις αρχές. Και με χαρά θα σας ε, βοηθήσουμε στην προετοιμασία σας με όποιο τρόπο μπορούμε. Αλλά ήδη και εδώ σημαντικό εργαλείο είναι η εκθέση ΑΝΑΝ. Αλλά να μην ξεχνάμε, η επίσκεψή σας στα μέσα Φεβρουαρίου θα είναι πολύ σημαντική για μας. επίσης προσβλημάτων. Αυτό λοιπόν αποτελεί μια επιπλέον ευκαιρία προβολής. Ε. Η κυρία Ντέιλι, τώρα και η Λία Ρέτσα έχει το λόγο. Μάλιστα, ευχαριστώ. Να απαντήσω στο ερώτημα της κυρίας Μούντι, η οποία μεν έφυγε, αλλά έχω κάτι να σχολιάσω και την λύση που έχει ακολουθηθεί, στην Ιορδανία, στο Λίβανο, όπου έχει γίνει υποδοχή τεράστιο εξέλιξη και αναπτύξη σε κάποιου μήνε στο Κοινοβούλιο. Θα υπάρχει και ενδιάμεση αναθεώρηση, και σχετική μάλλον συζήτηση για την ενδιάμεση αναθεώρηση. Ελπίζουμε να συνεχίσει. Είναι απαραίτητο να υποστηρίξει τον Μπαγκλαντέ και θα πρέπει να το ζητήσει αυτό τον Μπαγκλαντέ. Η άποψή του επί του παρόντο είναι ότι η Ροχίνγκα. Σύμφωνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνάδελφοι, δεν ξέρω αν έχετε περαιτέρω σχόλια και ερωτήματα. Ας ξεκινήσουμε σε 5 λεπτά παρακαλώ. Ladies Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να συνεχίσουμε με τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Περνάμε λοιπόν στο σημείο υπαριθμών 13, δηλαδή ανταλλαγή απόψεων με τον επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικής Πολιτικής και Εθνική ασφάλεια τη Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή του Ιράν. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Αλαντίν Μπουρουτζέντη που παρευρίσκεται στην ε, συνεδρίαση, τη σημερινή συνεδρίαση της ε, Επιτροπής μας. Ως επικεφαλής αυτής της Επιτροπής εθνικής ασφάλειας της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής ε, του Ιράν. Μπορείτε να μας ενημερώσετε σε σχέση με τις ε, εξελίξεις στη χώρα σας, ε, αλλά και τις αναταραχές που σημειώθηκαν εκεί, αλλά και να μας ενημερώσετε σε σχέση με το Comprehensive Plan of Action, το συνολικό δηλαδή σχέδιο δράσης για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Επιτρέψτε μου εμένα να κάνω κάποια εισαγωγικά σχόλια σε σχέση με αυτή τη συμφωνία την JCPOA. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να υποστηρίζει αυτή τη συμφωνία και παραμένει πλήρως δεσμευμένη σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της στο ακέραιο. Συζητήσαμε αυτό το ζήτημα και στην Ολομέλεια του Στρασβούργου την περασμένη εβδομάδα και εγώ παρακολούθησα τη συζήτηση που έγινε εκεί και διαπίστωσα πως όλες οι πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου παρά την δέσμευση που έχουμε αναλάβει σε ό,τι αφορά την συμφωνία αυτή, την JCPOA, άσχησαν επίσης κριτική ε, στο Ιράν και θεώρησαν πως θα πρέπει να σταματήσει την υποστήριξή της απέναντι στο καθεστώς του Ασάντ που ευθύνεται για απάνθρωπα εγκλήματα πολέμου στη Συρία. Ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν μια σημαντική πτυχή της σχέσης μας ε, με το Ιράν και τα μέλη της Επιτροπής μας ε, παρακολούθησαν προσεκτικά τις αναταραχές εκεί. Μας ανησυχεί η βία και η απαράδεκτη απώλεια ζώων στη χώρα σας και οι συνάδελφοι αξίωσαν την απελευθέρωση των διαφόρων κρατουμένων αλλά και την πάυση, τον τερματισμό των, της εκτέλεσης των θανατικών ποινών και θα θέλαμε να μας ενημερώσετε σε σχέση και με αυτά τα ζητήματα ως προς τη χώρα σας. Και κάτι ακόμα θα ήθελα να σας αναφέρω, κύριε Πρόεδρε. Εγώ είμαι Γερμανός και να σας πω ότι την περασμένη εβδομάδα οι δικές μας αστυνομικές αρχές προέβησαν σε κάποιες έρευνες 10 ατόμων ε, τα οποία, για τα οποία υπάρχουν υποψίες ε, πως δούλευαν ως πληροφοριοδότες μυστικοί δηλαδή πράκτορες του Ιράν. Υπάρχουν καταγγελίες λοιπόν για αυτά τα 10 άτομα ε, σε ό,τι αφορά ε, στόχους τρομοκρατικών επιθέσεων ε, εβραϊκών και Ισραηλινών γενικότερα, συμπεριλαμβανομένων για παράδειγμα εβραϊκών παιδικών σταθμών. Κάτι τέτοιο βέβαια μας δημιουργεί ιδιαίτερη ανησυχία. Οπότε αναμένουμε συνάδελφοι όλοι μας με μεγάλο ενδιαφέρον τη συζήτηση που θα κάνουμε σε σχέση με τις εξέλιξεις στη χώρα σας αλλά και α, τα, της εξωτερικής ε, πολιτικής σας. Θα θέλαμε λοιπόν να ακούσουμε την άποψή σας, κύριε Πρόεδρε, και έχετε το λόγο. Θα μιλήσει σε φάση ο κύριος ε, Πρόεδρος και όποιος θέλει να ακούσει απευθείας ε, την διαμήνα σε φάση ή κατευθείαν μάλλον τον ε, λόγο σε φάση. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ε, ευκαιρία να συμμετάσχω στην ε, σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής σας. Και παρευρίσκομαι σήμερα εδώ με κάποιους την πολύ καλή διοργάνωση αυτής της σημερινής συζήτησης αυτή τη συνάντηση και τον ευχαριστώ για την ευκαιρία που μα έδωσε σε όλου μα, του εκπροσώπου δηλαδή των χωρών μα, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις Ένωση απέναντι στη συνεργασία και τη διεύρυνση αυτής της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σημαντική. Ε, και αν δούμε ε, και την περίοδο πριν από, την, από το Σύμφωνο για τα Πυρηνικά υπήρχε κάποια ε, ένα πάγωμα, αν θέλετε, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της ε, οικονομικής μας ε, και πολιτική συνεργασίας των σχέσεων μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν δισεκατομμύρια δολάρια επενδύσει και πολιτικές ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων αλλά από εκεί και μετά ε, υπήρξαν πάρα πολλές κυρώσεις που επιβλήθηκαν αρχικά από τις ε, Ηνωμένε Πολιτείες λόγω δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι ουσιαστικά βρεθήκαμε σε μια απελπιστική θέση ε, γιατί ουσιαστικά υπήρξε αντίστοιχη αύξηση των εμπορικών μας σχέσεων με την Κίνα και με, κατά κάποιο τρόπο η βάση μετά τη σύναψη αυτού του πυρηνικού συμφώνου του JCPOA που αποτελεί βέβαια ένα κατακυρωμένο διεθνούς ε, κύρους ε, ε, σύμφωνο, ε, να πούμε ότι πραγματικά ε, έχει λάβει την έγκριση των Ηνωμένων Εθνών και δημιουργεί λοιπόν, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για αυτό το νέο κεφάλαιο, αυτή την ευκαιρία που μας δίνεται και βλέπουμε με χαρά να αυξάνονται πράγματι οι επαφές μας, οι διμερείς επαφές και σε οικονομικό επίπεδο και σε επιχειρηματικό αλλά και σε κοινοβουλευτικό. Αμέσως είδαμε και ποια είναι η, η, εικόνα που έχει ο πρόεδρος ε, Τραμπ ε, σε μια σειρά από ε, χώρες ανά τον κόσμο, όχι μόνο δηλαδή στο Ιράν και πώς φέρεται στην, σε διεθνές επίπεδο. Βλέπουμε δηλαδή ότι ουσιαστικά δεν συμμορφώνεται. Α, θεωρήσαμε Κάτι το ε, πολύ ε, παράξενο το ότι προέβη μια τέτοια προσβολή ε, ανθρώπων δηλαδή οι οποίοι απλά έχουν ένα διαφορετικό χρώμα. Και βέβαια είδαμε ποια ήταν η αντίδραση από εκεί και με τα σχόλια από την πλευρά ε, διαφόρων συνόντων. Αλλά είδαμε βέβαια και τα όσα είπε από εκεί και μετά ο πρόεδρο ε, Τραμπ σε σχέση με τη JCPOA, ότι δηλαδή ε, επιθυμεί να εγκαταλείψει την εφαρμογή αυτή τη συμφωνία, πράγμα βέβαια το οποίο ουσιαστικά θα υπονομεύσει τα όσα επιτύχαμε μέχρι τώρα. Και κάτι τέτοιο βέβαια αποτελεί, αφού προέβη ένα επίσημο ψήφισμα σε σχέση με αυτό το ζήτημα και επί τη βάση του οποίου ψηφίσματο εγκρίθηκε η πυρηνική συμφωνία JCPOA. Άρα λοιπόν αποτελεί προσβολή ναι και απέναντι στο Συμβούλιο Ασφαλεία των Ηνωμένων Εθνών. Εμεί όμω ε, θεωρούμε, εξακολουθούμε να θεωρούμε σημαντική αυτή τη συνεργασία. Εμεί ε, δεν επιθυμούμε ε, τη διάδοση. Υπάρχει ακριβώς υπάρχουν τέτοιου είδους ε, κανόνες, τέτοιου είδους ε, διατάξεις, ε, όμως βλέπουμε ότι δεν την χάνουν σεβασμού. Υπάρχουν δηλαδή άλλοι οι οποίοι προβαίνουν στην περαιτέρω έρευνα σε σχέση με τα πυρηνικά. Κάτα τον πόλεμο ο οποίος είχε αστηθεί κατά της χώρας μας είχαμε πάρα πολλές χιλιάδες αμάχων οι οποίοι ουσιαστικά βρέθηκαν θύματα χρήση ε, χημικών όπλων. Ε, και πραγματικά έχουμε ακόμα χιλιάδε πολίτε μα οι οποίοι εξακολουθούν κον όπλων. ουσιαστικά είχε μεταφερθεί η σχετική τεχνογνωσία από ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ε, εκεί. Οπότε και εμείς είχαμε για παράδειγμα εξετάσει επανειλημμένα πυράβλους οι οποίοι είχαν εκτοξευθεί κατά τη χώρα μας σε διάφορα 68 παιδιά έχασαν τη ζωή του στο πλαίσιο αυτής της επίθεση. και εμείς σε αυτό το πλαίσιο δεν είχαμε τη δυνατότητα να αμυνθούμε ακόμα και όταν χρησιμοποιήθηκαν ε, κατά του Ιράν χημικά και βιολογικά όπλα. Αλλά λοιπόν ε, σας καλούμε να ε, κρίνετε εσείς οι ίδιοι τη βασική αρχή για μια σταθερή ασφάλεια μιας χώρας. Το ότι λοιπόν εμεί ακολουθούμε τι δικέ μα αμυντικέ πολιτικέ δεν σημαίνει ότι προσπαθούμε να προσβάλλουμε την κυριαρχία άλλη χώρα. Θέλουμε ε, σχέσει καλή γειτονία. Έχουμε και τι κατάλληλε ικανότητε σε αμυντικό επίπεδο. Ε, και γι' αυτό έχει ε, επανειλημμένα βέβαια τεθεί και το σχετικό ερώτημα για το Ιράν. Γιατί δηλαδή επιθυμούσε ε, τα πυρηνικά όπλα. Η Σαουδική Αραβία, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ε, εδώ και τρία χρόνια βομβαρδίζει 800.000 άτομα ε, αυτή την περίοδο ε, υποφέρουν από χολέρα και από τις ε, θανατηφόρες βέβαια επιπτώσεις ε, αυτής της ασθένειας. Πέραν των όσων θυμάτων δηλαδή χάνουν τη ζωή τους από αυτές τις επιθέσεις, τα νοσοκομεία έχουν γεμίσει από παιδιά και εδώ βλέπω την διαξαγωγή πολέμου. Άρα λοιπόν τι είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, απλώς κάποια ωραία λόγια. Τι έκανε το ε, ε, Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Η Εμένη, για παράδειγμα, έχει καταδικαστεί ενώπιον ε, του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά διθέτως η Σαουδική θύματα. Και ε, πώς το κατάφερε αυτό η Σαουδική Αραβία μέσω ακριβώς ε, χρημάτων τα οποία δαπάνησε ουσιαστικά με αποτέλεσμα να σιωπήσουν κάποιοι και να μην αναφερθούν σε κάτι παραπάνω. Άρα λοιπόν πώς με αυτόν τον τρόπο πραγματικά ορίζονται τα δικαιώματα των παιδιών, τα δικαιώματα των γυναικών. Θα σα αναφερθώ και στην στα εσωτερικά της χώρας μας. Αλλά σε σχέση με τη Συρία ε, θα πρέπει να πω κάτι σημαντικό. Δεκάδες χιλιάδες τρομοκράτες εκπαιδεύτηκαν και έλαβαν χρήματα αλλά ανατρέψουν την κυβέρνηση και να υπάρξει αλλαγή του καθεστώτος. Αλλά ποιο ήταν το τελικό αποτέλεσμα. Δεκάδες χιλιάδες άμαχοι έπεσαν θύματα αυτής της ε, διαμάχης ε, και έχασαν τα σπίτια τους βλέπουμε όλους αυτούς τους ε, πρόσφυγες ε, και ε, υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Εμείς εδώ και 35 χρόνια φιλοξενούμε 3 εκατομμύρια Αφγανούς οι οποίοι βρέθηκαν εκτός Αφγανιστάν ακριβώς λόγω του πολέμου. Και εκατοντάδες χιλιάδες Αφγανοί λαμβάνουν εκπαίδευση, είναι απόφοιτοι ιρανικών πανεπιστημίων. Και ε, βέβαια όλα αυτά σας τα λέω γιατί ε, ε, υπάρχει και ένα σοβαρό πρόβλημα ανεργία σήμερα στη χώρα μας γιατί έχουμε όλους αυτούς τους Αφγανούς οι οποίοι η παρέμβησή μας ήταν ίδια. Δεν θέλαμε εμείς να παρέμβουμε στη Συρία για να παρισφρήσουμε στα, στις εσωτερικές υποθέσεις της Συρίας. Όχι, θέλαμε να υποστηρίξουμε αυτή τη χώρα ούτω ώστε να αντιμετωπίσουμε το ISIS που είναι η πιο επικίνδυνη θα υπήρχε, ε, δεν θα υπήρχε Συρία ω χώρα τη σήμερα ε, μέρα θα υπήρχε μια αναρχία, θα υπήρχε το απόλυτο χάο στην ευρύτερη περιοχή. Νομίζετε για παράδειγμα πως η κατάσταση στη Λιβύη τη σήμερα ημέρα είναι ικανοποιητική. Όχι. Αλλά πού οφείλεται αυτή η κατάσταση στη Λιβύη, στα όσα έκανε το ΝΑΤΟ και στο γεγονός ότι δεν ήταν σε θέση να ελέγξει τη συνέχεια ε, ε, της του ΕΕΤ. Άρα λοιπόν ε, το ίδιο δεν συνέβη ε, στη Συρία. Και αυτό οφείλεται ακριβώ και στη δική μας ε, παρέμβαση. Και, και βέβαια αυτό ισχύει και για τον Λίβανο. Ο Λίβανο είναι ένα μικρή, σε ένα εξάγει πολύ περισσότερη τρομοκρατία το ISIS προ την Ευρώπη. Ε, κατά του αρχικού μήνε τη κρίση στη Συρία, γιατί βρισκόμαστε βέβαια ήδη στο 7ο έτο τη κρίση στη Συρία, εμεί βρεθήκαμε σε ε, επαφή με ε, εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, έγιναν συναντήσει και με μένα προσωπικά και με τη δική μα βούλα. Τι είδατε όμω τελικά να συμβαίνει ότι πράγματι χιλιάδες ε, πολίτες και γυναίκες μάλιστα έχουν ε, ε, χώρες τους. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν εκπαιδευτεί ως τρομοκράτες, θα αποτελούν δηλαδή σημαντικό κίνδυνο για αυτές τις χώρες. Οι υπηρεσίες πληροφοριών μας λοιπόν έχουν κάποια εκτεκτικά και θα τα βάλουν σε ένα φορτηγό και θα κατευθυνθούν σε ένα κτίριο. Άρα λοιπόν θεωρούμε πως όταν υπάρχει τρομοκρατία τότε δεν πρέπει να δείχνουμε κανένας είδου σύκτο, η οποία έχει οδηγήσει σε 17.000 θύματα είναι τρομοκρατική οργάνωση. Απλά επειδή δηλαδή αλλάζει ε, ονομασία, ξαφνικά ε, διαδηλώσει οι οποίε ε, λαμβάνουν χώρα. Και πράγματι στη δική μα περίπτωση υπήρξε αυτή η βία διαδήλωση. Οι αστυνομικέ αρχέ χρειάστηκε να παρεύουν. Αλλά το Και στη δική μας στη Συμβουλευτική Επιτροπή υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι διαφωνούν μαζί μας, οι οποίοι εκφράζουν αντίθετες απόψεις και οι οποίοι εκφράζουν τα παραπονά τους. Αυτά είναι όλα αποδεκτά. Αλλά αν από εκεί και μετά ε, υπερβούν κάποια συγκεκριμένα όρια, όρια ασφαλείας, προφανώ και θα χρειαστεί να επέμβουν οι αστυνομικέ αρχέ. Αυτό ισχύει σε όλε τι χώρε του κόσμου. Στο Βέλγιο, για παράδειγμα, αν συμβεί κάτι τέτοιο, αυτά τα άτομα θα τεθούν υποκράτηση. Το ίδιο λοιπόν ισχύει στο Ιράν. Όσο ε, έλαμβαναν χώρα διαδηλώσει, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Όταν όμω αρχίσαν να πυρπολούν ε, ε, ή να επιτίθενται σε στρατιωτικέ εγκαταστάσει, προφανώ χρειάστηκε να επέμβουμε κι εμεί. Αυτό το είδαμε σε όλες τις χώρες και στο Βέλγιο πριν ε, μεταβώ. Ε, ρώτησα πώς είναι πολιτική πολιτική Αυτό το ρώτησα πριν ε, μεταβώ στο Βέλγιο. Μου είπαν ότι είναι 18. Όταν γυρίσω ε, μπορεί να είναι διαφορετικός ο αριθμός Δεν έχουμε διαφορετικά πρότυπα ανάλογα με τη χώρα. Υπάρχει ελευθερία του συνέρχεστε, του συνεταιρίζεστε, ε, υπάρχει ελευθερία για ε, διαδηλώσεις, αλλά υπάρχουν και κόκκινες γραμμές. Αυτή τώρα που μιλάνε για κατασκόπους, ε, θα γνωρίζετε ότι στο Ιράν έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που έχουν διπλή υπηκότητα. Μπορούν να βρίσκονται στην Ευρώπη, στον Καναδά και οπουδήποτε αλλού. Αν δείτε το σύνταγμά μας, βλέπετε όμως ότι όποιος αποκτήσει άλλη υπηκότητα χάνει την Ιρανική. Δυστυχώς όμως ε, μεταβαίνουν εκ νέου στο Ιράν για να δούνε την οικογένειά τους. Αλλά αυτό δεν πρέπει να το συγχέουμε με την κατασκοπία. Ο Αλτζαλή ε, είχε πανεπιστημιακή μόρφωση ήρθε στις στρατιωτικές μας εγκαταστάσεις και μετέφερε πληροφορίες. Και στη συνέχεια δύο πυρηνικοί μας επιστήμονες δολοφονήθηκαν. Και στη συνέχεια κάλεσε Ευρωπαίους και τους διέθεσε συγκεκριμένα φιλμ για κατασκοπία και ούτω καθεξής. Ο χρόνος μου είναι πολύ περιορισμένος και κάτι άλλο. Και στις είπα, όπως είπα στην αρχή, μπορεί να δεις. Έχουμε και πιο στενές σχέσεις στο μέλλον. Mr. Ευχαριστούμε για τα καλά. Να καλωσορίσω τον κύριο Μοχαμάτ Μπάνι Μουραμάτι και τον κύριο Χάντι Σουστάρη που είναι μέλη του Ιρανικού Κοινοβουλίου και φυσικά και τον πρέσβη του Ιράν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ώρα μέχρι τις 12.30 ίσως θα ήθελα να περιοριστούν οι ομιλητές στα δύο λεπτά. Ζητώ συγγνώμη, ξέρω πόσοι είναι ομιλητές, θα προσπαθήσω να δώσω το λόγο σε όλους. Ο κύριος Σαλαφρά ήθελα να χαιρετήσω τον πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Ισλαμικής ε, προηγούμενη εβδομάδα και πριν από την ε, επίσκεψη της ΑΦΕΤ στη χώρα σας, ο χρονισμός αυτός λοιπόν της δικής σας επίσκεψης είναι πολύ καλός. Το θέμα της συμφωνίας για τα πυρηνικά στο Ιράν είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, διότι υπάρχει θέμα κλιμάκωσης. Υπήρχε θέμα κλιμάκωσης, αλλά ο Διεθνός Οργανισμός, ο Διεθνής Οργανισμός Πυρηνικών Όπλων ε, θεωρεί ότι πληρούνται οι όροι συμμόρφωσης από το Ιράν. Θα πρέπει να δούμε φυσικά και το θέμα των ανθρωπιστικών δικαιωμάτων. Να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί στη χώρα σας και γιατί είχαμε τόσους ε, θανάτους και η ΕΠΑ ε, εξέφρασε τις ανησυχίες μέσα στα πλαίσια της συμφωνίας, εξέφρασε ανησυχία για την ε, πολιτοφυλακή σας και την μετάβαση μέρους της πολιτοφυλακής σας στη Συρία. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε ποιες είναι οι δικές σας αντιδράσεις σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα σας, διότι εμείς καταδικάζουμε τη θανατική ποινή που υπάρχει στη χώρα σας και να μας πείτε τι σκέφτεστε, τι επί της θανατικής ποινής. Ευχαριστούμε κύριε Σαλαφράγκα. Ο κύριος Φλέκενστάιν από τους Δημοκράτες και Σοσιαλιστές. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, και από το Ιράν θα συνεχιστούν οι συζητήσει. Είναι σωστή η χρονική συγκυρία και η πυρηνική συμφωνία τι δημιουργεί πιο πολύ εμπιστοσύνη και γι' αυτό λοιπόν έχει έρθει η στιγμή όχι να μιλάμε πλέον αλλά να εφαρμόσουμε τα δικά μας, αυτό που μας αναλογεί. Και είναι σωστή να διευκολυνθούν τέτοιες συζητήσεις επικοδομητικές, ειλικρινείς, με αμοιβαίο αλληλοσεβασμό. Και γι' αυτό λοιπόν ε, το πυραυλικό. Και σε ό,τι αφορά τη συμπερίληψη μόνο ενό τμήματο των φορέων, των εμπλεκόμενων φορέων, θεωρώ ότι ευνοεί αυτούς που δεν δεσμεύονται από τις λύσεις αυτές ε, και γι' αυτό λοιπόν ε, ανακύπτουν πολλά ζητήματα σε ό,τι αφορά την πολιτική της χώρας σας αλλά και άλλων χωρών της περιοχή Και ασφαλώς και θεωρούμε ότι το κοινοβουλίο αυτό και το έχει πει μάλλον πάντα με αυτά τα οποία δηλώνει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργό, αλλά το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ θεωρώ ότι δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αμφισβητηθεί. Θα πρέπει στο σημείο αυτό να κλείσω, αλλά θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να ανταλλάξουμε απόψεις για να υπάρξει καλύτερη κατανόηση. Ευχαριστούμε κύριε Φλέκενσταν και τώρα για το ECR το λόγο έχει ο κύριος Μπέλντερ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. να ε, αύριο ε, θα έχουμε την επέτειο του λοκαυτώματος. Ως ιστορικός είμαι άναυτος με το φαινόμενο του τε σε μια τέτοια συζήτηση και σας το θέτω αυτό το ερώτημα άμεσα. Ύστερα, διαμαρτυρών σε ό,τι αφορά τους ε, Ιρανούς νέους, σε ό,τι αφορά τους ε, Ιρανούς νέους. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής από την Άλντε, ο κύριος Αστρεβίτσιος. Διατεθμένος να απαντήσετε στις ερωτήσεις μας. Είμαι μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όπως ξέρετε, το Ιράν έχει το υψηλότερο ποσοστό θανάτωσης, κατά κεφαλή θανάτωσης στον κόσμο. Ε, κύριε Μπουρουζέρντι, γύρω υψηλά. Αύριο η Ευρώπη και ο ελεύθερος κόσμος ε, θα ε, τιμήσουν το ολοκαύτωμα είναι ένα ε, ιδεχθές ε, παράπτωμα και έγκλημα κατά της ανθρωπίνης. Ε, ακριβώς να τιμήσουμε αυτή την ημερομηνία. Η κυρία Σακοράφα έχει το λόγο για δύο λεπτά. Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κύριε Πρόεδρε στην Επιτροπή μας. Δεν θα αναφερθώ στα θέματα της πυρηνικής συμφωνίας γιατί το έχω τονίσει επανειλημμένα. Η πυρηνική συμφωνία ισχύει και όπως μας διαβεβαιώνει ο Οργανισμός Πυρηνικής Ενέργειας εφαρμόζεται στο ακέραιο. Επομένως, το Κοινοβούλιο δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να συνδράμει όσες και εμένα δυναμητίζουν τη συμφωνία αυτή για λόγους είτε γεωπολιτικής είτε πολιτικής σκοπιμότητας. Όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι θέσεις μας δεν έχουν αλλάξει από το ψήφισμα που υιοθετήθηκε πρόπερση από την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου για τις μελλοντικέ σχέσεις Ιράν και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως θα σας θέσω τρία ζητήματα. Σε αυτά θα ήθελα να σταθώ. Το πρώτο αφορά στο εσωτερικό και έχει να κάνει και κοινωνικέ διεκδικήσει και για τα οποία ο, κύριος, ο πρόεδρο, ο κύριο Σουχανή, εξ αρχή αναγνώρισε το δικαίωμα στο λαό να, τα, να, να το έχει και να διαμαρτύρεται. Θα είχε επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το σώμα αν θα μπορούσατε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις καταγγελίες που αφορούν στην εμπλοκή στις διαδηλώσεις και τη σύλληψη πρακτών για της Αστάνα. Ε, την, ε, θα ήθελα να μου επισημάνετε ε, τη θέση σας σε σχέση με την τουρκική κυβέρνηση και την επιχείρηση που κάνει αυτή τη στιγμή στο καντόνι του Αφρίν και στην πόλη Μάμπιτς. Τέλος, Μάνπιτς. Τέλο, θα ήθελα να μου ξεκαθαρίσετε ποιο ρόλο βλέπετε να διαδραματίζει το Ιράν στο Παλαιστινίο. Γνωρίζουμε ότι το Ιράν έχει πάρει ξεκάθαρη θέση για την, κατά τη απόφαση του κ. Τραμπ να μεταφέρει την Αμερικάνικη πρεσβεία στα Ιεροσόλυμα. Και επίση, με δεδομένη την οξυμένη κατάσταση των σχέσεων με τη Σαουδική Αραβία, να μα πείτε σε ποιο βαθμό το Ιράν προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλίε για τη δημιουργία ενό συνασπισμού κοινού μετόπου με τα αραβικά κράτη. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Σακοράφα και ο κύριος Κάρβερ τώρα έχει το λόγο από το EFTP. Ευχαριστώ πολύ. Στο, ε, στην ε, Ιεμένη. Ο Χέλμαρ Μπρόκ από το ΕΛ. Περνάμε στο δεύτερο γύρο. Ε, εφόσον δηλαδή το Ιράν συνεχίσει να εφαρμόζει αυτή τη συμφωνία και αυτό το επιβεβαιώνει και Διεθνή οργανισμός ατομικής ενέργειας τότε και εμεί την περίπτωση της Βορειοκορέα. Μετά το δεύτερο επίπεδο, είναι η ανάγκη δράσης κατά του Ισλαμικού κράτους, του ISIS, αλλά πολέμου για την προσώπων, το proxy war δηλαδή. Και βέβαια αυτό το λέω και στους προσώπους της Σαουδικής Αραβίας, όπως το λέω και σε εσά. Δεν θα πρέπει δηλαδή από αυτή τη διαδικασία της ε, αναγνώριση του δικαιώματος ύπαρξης του Ισραήλ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο των Λόπε τώρα για του σοσιαλιστέ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και τους καλεσμένους μας που παρευρέθηκαν όπως έκανα πολλοί συνάδελφοι καθώς και ο Πρόεδρος την, ε, το γεγονός ότι θα συμβαδίσουμε με την εφαρμογή για τα πυρηνικά στο Ιράν και τη ευρύτερη περιφέρεια. Θα πρέπει όμως να μιλήσουμε για τα πρόσφατα γεγονότα στη χώρα σας που παρακολουθήσαμε με ενδιαφέρον αλλά και με ανησυχία σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και τη σταθερότητα της χώρας. Και θα ήθελα να επαναστατική πολιτική το φύλακι θα αναλάβει συγκεκριμένη όχι μόνο πολιτική αλλά και οικονομική δραστηριότητα και όσον αφορά τη θανατική ποινή και επίσης έγινε αναφορά και για τους διακινητές ναρκωτικών. Τρίτον, Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να σταματήσουν για έναν διάλογο σε περιφερειακό επίπεδο, τον οποίο προσ... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ. Ναι και η υποστηρίξη του Ιράν προς τη Χεσμολά. Το Ιράν φυσικά και θέλει να τη και νομίζω ότι μακροπρόθεσμα οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ιράν θα μπορούσαν να βελτιωθούν εάν το σχέσεις βολάχα. Ευχαριστώ. Είμαι ιδιαίτερα επικριτικός ως προς την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν και αυτό με την κατάσταση στην περιφέρεια δεν θα μπορούσε να υπάρχει μία συμφωνία χωρίς το Ιράν. Και υπ' αυτή την έννοια, αλλά αν δεν υπήρχε η Χεσμολά, αυτή τη στιγμή το Ισλαμικό κράτος θα ήταν μέσα στο Λίβανο. Αυτό, αλλά αν δεν υπήρχε η Χεσμολά, αυτή τη στιγμή το Ισλαμικό κράτος θα ήταν μέσα στο Λίβανο. Αυτό τη στιγμή που υποστηρίζεται ο γενοκτόνος ε, πρόεδρος της Συρίας, στην ουσία δεν μπορεί να οδηγήσει στην ειρήνευση στην περιοχή. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι το Ισλαμικό κράτος θα μπορούσε να έχει βρεθεί μέχρι τη Βαγδάτη. Γι' αυτό ο ε, στρατάχης Σουλεϊμάν ακολούθησε πολύ καλή τακτική γιατί αυτό που μας έμποτα δεν έχετε ούτε στρατιωτική παρουσία ούτε τη δυνατότητα να βοηθήσετε την ε, πολιτοφυλακή του Αλσαλαλάχ. Αυτή είναι μία απτή πραγματικότητα. Σας ευχαριστούμε Κρινάρτ και τώρα περνάμε στους τελευταίους τρεις εμερητές, σύμφωνα με τη λίστα, ο κύριος Ρεντάκτουσον είναι ο πρώτος. Thank uh, Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Μπουρουτζέρτη. Όπως δήλωσε και ο Πρόεδρος, ο κ. Μακάλιστερ, από την αρχή της συνεδρίασης, στην Επιτροπή μας ανησυχούμε. Ανησυχούμε βαθύτατα σε ό,τι αφορά τις τρέχουσε εξελίξει στη χώρα σα. Και πέραν τούτου η χρηματοδότηση της Ισμολάς, της Χαμάς, συμβάλλει στις πολλώσεις, την αστάθεια στις περιοχές και απειλεί την ασφάλεια του Ισραήλ, της μοναδικής δημοκρατίας, της Παϊκής Ένωσης. Είναι τόσο σημαντικές για σας. Σας ρωτώ, με τι τρόπο εισακούεται τι ανησυχίε και την κριτική από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση τη τρομοκρατία. Δεύτερη ερώτηση. Είστε πρόεδρο συνέλευση. Ξέρουμε ότι στις πρόσφατες διαδηλώσει. μα, πάνω από 3.000 άτομα, 3.700 άτομα. Συζητήσαμε την ε, νεαρών διαδηλωτών οι οποίοι θανατώθηκαν μετά από βασανίστηρια, μετά την έναρξη των ε, φαινομένων αυτών. Και σας ρωτώ λοιπόν, ε, σε τι βαθμό είστε υπεύθυνοι και τι κάνετε για να απελευθερωθούν, ε, κυρία Μπουρούτζερδη. Πιστεύω ότι η Πρινική Συμφωνία αποτελεί μια μεγάλη λύση ό,τι αφορά την περιφερειακή, τον περιφερειακό αντίκτυπο που θα είχε εμβάθυνση των σχέσεών μας και είναι, είναι η εναλλακτική για την επιδείνωση της ε, περίπτωσης της Βορείου Κορέα. Ό,τι καλύτερα μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε την ε, περαιτέρω επέκταση. Με την ευκαιρία λοιπόν αυτή, κατά δεύτερον, στο μέλλον, στο μέλλον, όχι τώρα, πώς θεωρείτε ότι θα διαμορφωθούν οι σχέσεις σας με το Ισραήλ και πώς θα είναι οι μελλοντικέ σας σχέσεις με την Σαουδική Αραβία. Γιατί το Ιράν και η Σαουδική Αραβία αποτελούν μια ενδυναμή λύση και ευκαιρία της σταθερότητας. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμα πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της. Ήταν μέχρι τώρα μια ελεύθερη χώρα. Κατάγεστε από μια χώρα με πολύ σημαντικά πολιτιστικά μνημεία και εβδομάδες ε, με την βία καταστολή των ε, διαδηλώσεων στη χώρα σας. Ε. Οπότε θα ήθελα εδώ να σας ρωτήσω πώς διασφαλίσετε την ανθρώπινη μεταχείριση αυτών των κρατούμενων ε, και πώς θα διασφαλίσετε την απελευθέρωσή τους ε, και πώς θα εγγυηθείτε το λόγο στον πρόεδρο της... Ε, κύριε Πρόεδρε, προσπαθήστε να συνοψίσετε σε 10 λεπτά τις απαντήσεις σας, γιατί θα έχουμε πρόβλημα από εκεί και μετά με τη διερμηνία αν καθυστερήσετε παραπάνω ένα ερώτημα από τη δική μου πλευρά. Η αληθεύει αυτή η κατηγορία που αναφέρθηκε ότι πράγματι υπήρξαν δηλαδή κατάσκοποι της δικής σας ε, χώρας οι οποίοι στη Γερμανία προσπαθούσαν να εντοπίσουν κάποιους τρομοκρατικούς ε, στόχους ε, συμπεριλαμβανομένων και παιδικών σταθμών. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αν ήξερα ότι θα μου τεθούν τόσα πολλά ερωτήματα, θα είχα προσέλθει νωρίτερα, γιατί πραγματικά θέλω πάρα πολύ να προβούμε σε ανταλλαγή απόψεων. Και οι δύο πλευρέ ε, είμαστε εκπρόσωποι των πολιτών μα, των λαών μα. Ε, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο στι απαντήσει μου, ακριβώ επειδή μου είπατε ότι έχω περιορισμένο χρόνο. Καταρχήν θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για την υποστήριξή σας απέναντι στο την ολοκληρωμένο σχέδιο δράση το JCPOA, το πυρηνικό δηλαδή σύμφωνο, και τα σχετικά ερωτήματα ε, που τέθηκαν ε, από εκεί και μετά ε, ουσιαστικά ήταν κοινά από διαφόρους συναδέλφους οπότε θα αναφερθώ από κοινού σε αυτά. Τέθηκαν πολλά ερωτήματα σε ό,τι αφορά τις διαδηλώσεις στη χώρα μου, σε ό,τι αφορά το Ισραήλ, σε ό,τι αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άρα δεν θα απαντήσω σε κάθε βουλευτή ξεχωριστά. Θα δώσω απαντήσεις για τα ίδια θέματα σε όλους. Ε, να σας πω ότι οι αστυνομικοί, για παράδειγμα, στη χώρα μας δεν φέρουν όπλα. Αντιθέτως, για παράδειγμα, στον Καναδά ή στις ΗΠΑ έχουν το δικαίωμα ακόμα και οι τροχονόμοι να οπλοφορούν. Ε, πρόσφατα, για παράδειγμα, στον Καναδά υπήρχε άσκηση βίας και έχασε τη ζωή του ένας ε, πεζός από το Αντιθέτω, λοιπόν, στη δική μα χώρα υπάρχει αυτοσυγκράτηση από την πλευρά των αστυνομικών, οι οποίοι δεν οπλοφορούν, επαναλαμβάνω, ε, και επέδειξαν αυτή την αυτοσυγκράτηση απέναντι στου διαδηλωτέ. Και υπήρξαν δεκάδε, για να μην πω εκατοντάδε, από αστυνομικού οι οποίοι τραυματίστηκαν, ε, χωρί ε, να αντιμετωπίσουμε το ίδιο τρόπο αυτού του διαδηλωτέ. Και μπορώ να σα δώσω αντίστοιχα παραδείγματα για το τι έχει συμβεί στο Βέλγιο, στη Γερμανία, στη Γαλλία και αλλού. Όπου δηλαδή ε, υπερβαίνει αν θέλετε κάποιες κόκκινες γραμμές ασφαλείας, ε, τότε προφανώς αναλαμβάνει δράση το κράτος. Και εγώ δεν είπα ότι όσοι έχουν τεθεί υποκράτηση θα παραμείνουν ε, σε βάθος χρόνου υποκράτηση. Ήδη σήμερα, για παράδειγμα, σε ε, επικοινωνία που είχαμε τον ε, επικεφαλής εκεί του συμφωνιστικού καταστήματος υπήρξαν ε, και άλλοι οι οποίοι απελευθερώθηκαν. Οπότε πραγματικά ας μην υπερβάλλεται. Δηλαδή υπάρχει πραγματικά το δικαίωμα διαδήλωσης στο Ιράν και χαίρουν αυτού του δικαιώματος οι πολίτες μας εφόσον, επαναλαμβάνω, δεν υπερβαίνουν κάποια όρια, εφόσον δεν βάζουν φωτιά σε κτίρια ε, και δεν προβαίνουν σε βανταλισμούς. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πυρηνικό σύμφωνο, Μα είπατε πω είναι σημαντικό αυτό το σύμφωνο και από εκεί και μετά σα λέω σε ό,τι αφορά του πυραυλού, αυτό είναι το μηνωτικό μοναδικό όπλο που έχουμε στη διάθεσή μα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στο μέλλον κάποιο όπω ο Σαντάμ να επιτεθεί στη χώρα μα, χωρί εμεί να μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ποιο είναι ο ρόλο, ποια είναι η υποχρέωση των ενόπλων δυνάμεών μα. Να έχουμε τη δυνατότητα να αμυνθούμε. Δεν θέλουμε να έχουμε τα όπλα που έχουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Δεν έχουμε δηλαδή ε, όπλα μαζικής καταστροφής και είμαστε κατά της χρήσης τέτοιων όπλων μαζικών. Αλλά από την άλλη πλευρά ε, αντιληφθείτε ότι προφανώς χρειάζεται να έχουμε κάποια όπλα, κάποιε ένοπλε ικανότητε, αμυντικές ικανότητε, αποτρεπτικού χαρακτήρα έτσι ώστε, έτσι ώστε να μπορούμε να αμυνθούμε. Όχι για να απειλήσουμε κάποιον άλλον. Η Σαουδική Αραβία η οποία βρίσκεται ε, για παράδειγμα στην ίδια περιοχή έχουν ε, μεγαλύτερου βενιλοκού ε, πυράβλου και μάλιστα αυτέ τι μέρε προέβησαν σε αγορέ χιλιάδων περαιτέρω πυράβλων από την Κίνα. Άρα λοιπόν, το να μπορούμε να διαθέτουμε αυτού του πυράβλε είναι κάτι το αδιαπραγμάτευτο για μα και χρειαζόμαστε τέτοιου είδου ε, Απλώ Απλώς προσπαθώ να διευκρινίσω εδώ το γιατί χρειαζόμαστε τέτοιου είδου υπηρευλικά συστήματα. Ε, στην πρόσφατη επίσκεψη που έκανε ο πρόεδρο στράμψη στη Σαουδική Αραβία ε, έλαβε χώρα πώληση όπλων σε ύψο δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αλλά και άλλε χώρε του κόλπου δαπανούν πάρα πολύ υψηλά ποσά εκατοντάδε εκατομμυρίων ε, δολαρίων για τέτοιο είδου όπλα, ενώ άλλε χώρε τη ευρύτερη περιοχή διαθέτουν πυρηνικά όπλα. Άρα λοιπόν ε, ουσιαστικά εμεί προσπαθούμε να έχουμε την ελάχιστη αποτρεπτική αμυντική ικανότητα που χρειαζόμαστε, ακριβώ επειδή είμαστε θύμα και διαφόρων απειλών τι οποίε δεχόμαστε. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα τη Μέση Ανατολή γενικότερα. Ναι, ε, υπήρξαν μια σειρά από συμφωνίε του Όσλο, τη Μαδρίτη και τελικά δεν κατέληξαν πουθενά. Γιατί λέτε να συνέβη αυτό. Ε, το Ιράν ε, ε, παρενέβη στην εφαρμογή αυτών των συμφωνιών. Όχι. Γιατί λοιπόν δεν τελεσφόρησαν αυτές οι συμφωνίες. Το σιωνιστικό καθεστώς το οποίο δεν μπορούμε να αποδεχτούμε έτσι όπως δρά, ουσιαστικά έχουν προβεί σε κατάληψη της χώρας ενός άλλου λαού. Ουσιαστικά έχουν καταστήσει εκατομμύρια ανθρώπων άστεγου δεν, δεν, βρίσκονται στη χώρα τους και έχουν υπάρξει τόσα πολλά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών παρόλα αυτά το Ισραήλ δεν επιτρέπει σε αυτούς τους πρόσφυγες να επιστρέψουν ε, στην πατρίδα τους. Εμείς λοιπόν ως Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν λέμε ότι οι Παλαιστίνοι θα πρέπει να μπορούν να κάνουν ένα δημοψήφισμα για να επιλέξουν το καθεστώς το οποίο θα ισχύει για τους ίδιους. Και εμείς θα δεχτούμε οποιοδήποτε αποτέλεσμα θα προκύψει από ένα τέτοιο δημοψήφισμα. Αυτή τη στιγμή μόνο το 2% αυτής της περιοχής ανήκει στους ε, Παλαιστινίους. Ε, ε, και βέβαια όχι, και αυτό το 2% βλέπετε τι, τι σημαίνει για αυτούς. Τίθεται υποκράτηση, σκοτώνονται και διαβιούν υπό απελπιστικές συνθήκες. Και οι υπόλοιπε περιοχέ που βρίσκονται υπό την κατοχή του Ισραήλ, ουσιαστικά εκεί οι πολίτε ε, βρίσκονται ε, πραγματικά σε υποκράτηση αποκλεισμένη. Αυτό συμβαίνει. Δηλαδή σε πάρα πολύ μικρούς περιορισμένους θύλακες. Και ε, τα κάνει όλα αυτά το Ισραήλ και εσείς μας λέτε ότι παραβιάζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς καταρχήν έχουμε και θρησκευτικέ μειονότητες στη δική μας χώρα και η εβραϊκή μας κοινότητα στο Ιράν με βάση το σύνταγμά μας δικαιούται να έχει εκπροσώπους στην ε, Βουλή μας και το, το κάνει. Υπάρχουν τρεις εκπρόσωποι. Δύο από την, ε, από την αρμενική πλευρά και ε, έναν από, την, από τους Συρίους. Αλλά και εκπροσώποι του ζωραστρισμού εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο μας. Έχουμε λοιπόν αυτές τις εγγύσεις στο δικό μα ε, σύνταγμα. Υπάρχουν και εκκλησίε προφανώς. Και υπάρχουν και συναγωγές, εβραϊκέ συναγωγές. Ε, και ε, παλαιότερες τέτοιες συναγωγές ε, και εκκλησίες ανοικοδομούνται και ε, με δικά μας κονδύλια. Και από εκεί και μετά μας λέτε ότι παραβιάζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς έχουμε και γυναίκες οι οποίες ασκούν όλα τα επαγγέλματα. Είναι πιλότοι, οδηγεί τα πάντα. Και η Σαουδική Αραβία πρόσφατα επέτρεψε στις γυναίκες να μπορούν απλώς και μόνο να οδηγούν αυτοκίνητο. Και εσείς μας λέτε σε εμά ότι ως Ιράν έχουμε πρόβλημα με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, λοιπόν, όλοι είμαστε άνθρωποι. Κάποια στιγμή δηλαδή ερχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο και κάποια στιγμή καταλείπουμε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχει λοιπόν μια συνείδηση την οποία έχουμε. Ακόμα και αν δεν ε, πιστεύουμε στη θρησκεία και ακόμα δεν πιστεύουμε δηλαδή στη ζωή μετά θάνατον, σίγουρα έχουμε μια συνείδηση, ειδικότερα ως εκπρόσωποι, αξιότιμοι εκπρόσωποι των πολιτών μας. Εσείς λοιπόν ως εκπρόσωποι των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πώς αποδέχεστε ε, την, ε, το, το, ουσιαστικά τη θανάτωση χιλιάδων ε, αμάχων με ευθύνη της Σαουδικής Αραβίας. Γιατί δεν απευθύνεστε σε ένα ε, ποινικό δικαστήριο για, έτσι ώστε να στραφείτε κατά της Σαουδικής Αραβίας. Γιατί δεν το κάνετε, επειδή δηλαδή υπάρχουν κάποιε πολιτικές σκοπιμότητες από την πλευρά σας. Εκεί ξαφνικά σταματάνε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πραγματικά σα καλώ να εξετάσετε όλα τα ζητήματα με τον ίδιο τρόπο. Πρόκειται για ανθρώπινα ε, όντα σε όλες τις περιπτώσεις. Και δικός μας ο Μάμης είχε αναφέρει ότι όλα, όλοι οι άνθρωποι είναι άδελφοι μας. Είτε από θρησκευτική άποψη, είτε ως άνθρωποι. Γενικότερα. Έτσι λοιπόν όλοι μας έχουμε συνείδηση και γι' αυτό θα πρέπει να εξετάζουμε το σύνολο και να αντιμετωπίζουμε το σύνολο της ανθρωπότητας όλους ως ανθρώπινα όντα. Τώρα, αναφερθήκατε ε, στους φυλακισμένους ε, στο Ιράν. Χρήστες ναρκωτικών στη χώρα μας ε, και συχνά μας είπαν αυτοί οι λαθρέποροι ναρκωτικών ότι ουσιαστικά περνάμε από τη χώρα